Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des äh, Ausschusses für Haushaltskontrolle. Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σημείο 1 είναι η έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια, θεωρώ ότι είναι δεδομένη η έγκρισή σας για την ημερησία διάταξη δυνατότητες διερμηνίας, το έχετε και γραπτά στα έγκριτα Cont News. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρία αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο ζωντανή. Και φυσικά στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο Τη επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Μπορείτε να βρείτε όλα τα υγεία έγγραφα. Έρχομαι στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Δεν ε, ζητά κανείς το λόγο. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Έχουμε την ε, διαδικασία απαλλαγή και υπάρχει εδώ η εκπροσώπηση του Συμβουλίου και θα ήθελα να ζητήσω από την Υπουργό Εσωτερικών του ε, Βασιλείου της Δανίας, την κυρία Μαργκρέτε Βεστάκερ, να την χαιρετήσω για την παρουσία της στην Επιτροπή και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για να μας δώσει τις ε, θέσεις του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Εξάλλου είναι παρόν και ο κύριος Σεμέτα, ο αρμόδιος ε, επίτροπος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας και φυσικά και ο κύριος Φιέλνε ο εισηγητής για το θέμα αυτό θα λάβει στη συνέχεια το λόγο για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά εάν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο σημείο αυτό της ημέρας της διάταξης και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εμάς κυρία Βερστάκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά θα μιλήσω. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ε, προσβλέπω στο να προβάλλω το ρόλο του Συμβουλίου ακριβώς όπως προβάλλεται στο Συμβουλίο και αυτό σε σχέση με την αιτήσια απαλλαγή. Ε, Υπάρχει η σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την απαλλαγή τη Επιτροπής ως προς την εκτέλεση του προπολογισμού του 2010. Θα ήθελα λοιπόν να δράξω αυτή την ευκαιρία όχι μόνο για να σας παρουσιάσω τη σύσταση του Συμβουλίου που είναι ένα απαλλαγή επιτροπή, αλλά θα ήθελα παράλληλα και να επανεπιβεβαιώσω τη σημασία που αποδίδει το Συμβούλιο σε χρηστή οικονομική διαχείριση των Ταμείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελεγκτικό συνέδριο εφέτος ε, μας ε, έδωσε δύο μηνύματα, τα επισύναψε στην έκθεσή του. Πρώτον, εκφράζεται με σαφήνεια όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην εκτέλεση του προπολογισμού σε σχέση με προηγούμενα έτη. Το Συμβούλιο από τους ελέγχους και τα συμπεράσματα του συνεδρίου καταλήγει στο ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη κατά τα τελευταία έτη όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Αυτό αφορά τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη-μέλη. Διαπιστώνεται λοιπόν μια σταθεροποίηση. Ελήφθησαν ουσιαστικά μέτρα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αυτά απέδωσαν. Και αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, ένα μεγάλο κομμάτι των ε, ε, κονδυλίων ε, του προπολογισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων και η εποπτεία είναι μόνο εν μέρη αποτελεσματική ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων. Οι ιδιαίτερες αδυναμίες εμφανίζονται στη γεωργία, στους φυσικούς πόρους, Εκεί οι καταβολές ε, παρουσιάζουν ε, μεγάλο ποσοστό σφάλματος. Πρόβλημα υπάρχει και στη συνοχή, στην ενέργεια και στις μεταφορές. Και το ποσοστό σφάλματος αυξήθηκε σημαντικά σε 7,7% σε αντίθεση με την ουσιαστική βελτίωση που διαπιστώθηκε πέρυσι ε, στον τομέα της συνοχής. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο θετικό. Είναι σαφές ε, ότι ε, πόρο απέχουμε από τον στόχο μας που είναι να υπάρχει μία ε, γνώμη του Συμβουλίου άνευ επιφυλάξεων. Αυτό είναι ο στόχος. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την επιθυμία του ε, κάθε χρόνο να υπάρχει μείωση του ποσοστού σφάλματος και να υπάρξει και βελτίωση ε, στα διαχειριστικά συστήματα. Επίσης ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της όσον αφορά στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προπλογισμού, να ενισχύσει την εποπτεία και τον έλεγχο, τις σχετικές δομές και επίσης και να ενισχύσει τις συνεργασία της ε, με τις ε, εποπτικές αρχές των κρατών μελών. Ε, οι προσπάθειες που αφορούν στους κινδύνους της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων είναι απαραίτητες για να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος στις πληρωμές Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρχει η βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό προς όφελος βεβαίως των Ευρωπαίων πολιτών και των φορολογουμένων. Όλοι οφείλουμε να το γνωρίζουμε αυτό, κυρίως ε, τώρα που διερχόμεθα οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Η ιδιαίτερη σημασία αποζητείται στην σωστή εκταμείευση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω φέτος ε, ε, πρέπει να αποδοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή γιατί ε, σε τελική ανάλυση πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για το Συμβούλιο που αφορά στην ε, γνωμοδότηση άνευ επιφυλάξεων είναι η ε, συστηματική ο συστηματικό έλεγχο των πληρωμών, οποτεδήποτε υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ουσιαστικέ αδυναμίε στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Και αυτό μέχρι να εφαρμοστούν πλήρως διορθωτικές πράξεις. Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει τα λάθη που εντοπίζει χωρίς καθυστέρηση και αυτό με την ανάκληση των αχρεωστήτως ε, καταβλητέντων. Αυτό να γίνει μέσα από ε, οικονομικές διορθώσεις, ε, να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η εφαρμογή των διορθώσεων. Εξάλλου, το Συμβούλιο αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη σημασία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για την περίοδο την οποία εξτάζουμε. Παρ' αυτά, η τακτικές αξιολογήσεις της λειτουργίας είναι απαραίτητες για να εντοπίζονται αδυναμίες, όπως επίσης και δυνατότητες βελτίωσης η συνεχής αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών και οι διαπραγματεύσεις ε, στη σχετική νομοθεσία θα οδηγήσουν στο επόμενο πολιτές πλαίσιο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι σωστές και αποτελούν μια απαραίτητη ευκαιρία έτσι ώστε να υπάρξουν ε, χρήσιμες και κατάλληλες τροποποίησεις. Βεβαίως, η ισορροπία ανάμεσα στην προστιθέμενη αξία και το επιπρόσθετο διοικητικό ε, ε, και το ε, φορτίο του ελέγχου, αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί. Κυρίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά προγράμματα, ε, αυτό θα πρέπει να είναι το οδηγό νήμα για τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα. Ένα απλό σύστημα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόζεται από ένα περίπλοκο. Η πολυπλοκότητα των κανονισμών παραμένει ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί τα μάλα. Οι κανονισμοί πρέπει να καταστούν σαφέστεροι, περισσότερο συνεπείς, πολύ πιο εύκολοι στην εφαρμογή τους. Ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα, η οικονομική διαχείριση, ο, τομέας, ε, ο δημόσιος τομέας των αναθέσεων, σε αυτούς τους τομείς πρέπει να υπάρξουν απλουστεύσεις. Όπως και στο παρελθόν, ο τομέας των δημόσιων αναθέσεων και το 2010 ήταν ένας τομέας σημαντικών σφαλμάτων, κυρίως όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγξουν διεξοδικά και προσωπικά την νομοθεσία που αφορά στην, ε, σε αναθέσεις του δημόσιου τομέα, να δώσουν σημασία κυρίως στην αποτελεσματικότητα των κείμενων κανόνων και να ε, προσπαθήσουν στο μέλλον να λάβουν υπόψη τους ε, τις βελτιώσεις, αυτό να το εντάξουν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και για την οργάνωση των κανόνων σχετικά με τις αναθέσεις. Τώρα θα ήθελα να επανέλθω στι αντιναμίε που εντοπίστηκαν από το συνέδριο όσον αφορά στο εσωτερικό σύστημα ελέγχου τη Επιτροπή. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η, ο η ετήσια έκθεση ελέγχου που υποβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση, υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επιτροπή, βασίζεται στην αξιολόγηση των πόρων και στι διαδικασίε ελέγχου, που είναι χρήσιμα εργαλεία για να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων. Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο αποδίδει σημασία στο ότι η ε, τήσια έκθεση δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και πρέπει να είναι συγκρίσιμη έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η εσωτερική λογοδοσία, λογοδοσία μέσα στους ίδιους οργανισμούς. Γι' αυτό καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την συνεπή εφαρμογή των υποκείμενων πράξεων στις γενικές διευθύνσεις, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων που διεξάγει η Επιτροπή, με στόχο όπου είναι δυνατόν να διευρύνεται το φάσμα και η κλίμακα των ε, αποθεμάτων. Και τέλος, λόγω του ότι υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση όπου το συνέδριο παρουσιάζει την άποψή του για την αυτοαξιολόγηση της Επιτροπής ως προς την απόδοσή της ε, και επίσης και αξιολόγηση του συνεδρίου για την απόδοση της Επιτροπής. Αυτά έγιναν με βάση ειδικού ελέγχους και βάση ειδικέ εκθέσεις. Το Συμβούλιο επισημαίνει το πόσο σημαντικό είναι ε, να υπάρχει αποτελεσματικότητα στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον καθορισμό στόχων. Φαντάζομαι ότι Όλοι γνωρίζετε το ε, ακρονίμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο SMART, που είναι ε, Specific Measurable Achievement ε, and Time, είναι τα αρχικά στα αγγλικά SME το SMART, τον προηγούμενο μήνα το Συμβούλιο εξέτασε διεξοδικά τις λεπτομέρειες του προπολογισμού ε, της Επιτροπής για το 2010 με βάση τις επαρτήσεις που έκανε το συνέδριο στη δική του την έκθεση. Και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ για άλλη μια φορά υπενθύμησε σε όλου του άμεσα ενδιαφερόμενου και στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδο κατά τα επόμενα έτη. Ε, οι απόψει του Συμβουλίου οδήγησαν στη σύστασή του προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εγκρίθηκε ε, στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στι 21 Φεβρουαρίου να δοθεί απαλλαγή στην Επιτροπή ε, όσον αφορά στην εκτέλεση του προπολογισμού του 2010. Επίση, το Συμβούλιο ενέκρινε τι συστάσει για απαλλαγή των 22 οργανισμών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομική οντότητα και έλαβε ε, τις ε, προτάσεις τους που θα ενταχθούν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς μπορούν βέβαια να βελτιώσουν την διαχείριση των οικονομικών τους. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο συστήνει απαλλαγή για το σύνολο αυτών. Επιπλέον, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, το Συμβούλιο ενέκρινε συστάσεις να δοθεί απαλλαγή σε έξι εκτελεστικούς οργανισμούς και επτά ε, κοινέ επιχειρήσεις. Αυτές, αυτές είναι οι συστάσεις προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις που έγιναν, γιατί όπως σας είπα, ε, αυτά βασίζονται σε δύο συστάσεις. Η μία σύσταση είναι καλή, η άλλη λιγότερο καλή ε, και πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οτιδήποτε χρήση βελτίωσης πράγματι να το βελτιώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ, κυρία Βεστάγερ για την παρουσίαση που μας κάνατε από πλευράς του Συμβουλίου. Αν ε, δείτε τις συνθήκες και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν ε, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Οπότε οι συστάσεις σας όσον αφορά την απαλλαγή από πλευράς συστάσεις του Συμβουλίου δηλαδή είναι ένα σημαντικό θέμα για μας και εμεί, που είμαστε η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θεωρούμε ότι η διαδικασία απαλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς την Προεδρία της Δανίας για την διάθεση συνεργασίας που δείχνει το Συμβούλιο μαζί μας στο θέμα αυτό της απαλλαγής. Θέλω να το πω και να το τονίσω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας εδώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, αρχίζει η συζήτηση. Οπότε, το λόγο έχει πρώτα ο κύριος Φαλνε, που είναι και ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Υπουργό. Πρώτα απ' που ήρθατε εδώ. Χαίρομαι πολύ που βλέπω έναν εκπρόσωπο κράτους μέλους εδώ στην διαδικασία αυτή απαλλαγής, παρόλο βέβαια που βρισκόσαστε εδώ υπό την ιδιότητα της Προεδρίας του Συμβουλίου. Πάντως χαίρομαι πολύ. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της πολυπλοκότητας και της απλοποίησης. Είναι ένα θέμα που μπαίνει για πολλές επιτροπές, όχι μόνο για τη δικιά μας. Όμως αναρωτιέμαι σχετικά με τις ευθύνες που έχουμε εμείς από πλευρά των θεσμικών οργάνων. Δεν έχουμε εμείς την ευθύνη που η νομοθεσία είναι τελικά περίπλοκη και όχι απλοποιημένη. Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, την ευθύνη που έχουμε εμείς δηλαδή, στην νομοθετική αυτή διαδικασία. Πιστεύω πάντως ότι θα έπρεπε τα κράτη-μέλη, και ίσως εσείς θα μπορούσατε να το θέσετε αυτό στα κράτη-μέλη, να αναρωτηθούν και αυτά τελικά οι ευρωπαϊκές οδηγίες πώς μπορούν να φροντίσουν να τίθενται σε εφαρμογή όσο γίνεται πιο απλά. Εγώ γνωρίζω καλά τη Σουηδία, εσείς τη Δανία. Έχω όμως την αίσθηση ότι τα Υπουργεία των χωρών μελών έχουν αν μη τι άλλο την τάση κάθε φορά που θέτουν σε εφαρμογή μια νομοθεσία να προσθέτουν πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και τα οποία δεν έχουν απαραίτητα κάτι να κάνουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τις οδηγίες δηλαδή που εμείς ε, υιοθετούμε και που θα έπρεπε να τίθεται σε εφαρμογή στις χώρες μέλη. Και νομίζω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι όταν λέμε ότι τελικά στις εκλογικές μας περιφέρειες βρισκόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με τους πολίτες οι οποίοι λένε ότι φταίνε οι Βρυξέλλες κάθε φορά. Συνεπώ όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και θα ήθελα και εσείς να το μεταφέρετε αυτό στους συναδέρφους σας στο Συμβούλιο. Υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα που θέλω να μάθω από εσά. Αν δεν με πατάει μνήμη μου, στην τελευταία διαδικασία απαλλαγή, νομίζω υπήρχαν τέσσερις χώρες οι οποίες έστειλαν επιστολή, αν δεν απατώμε, Τρεις ή τέσσερις επίσης κράτησαν θέση αποχής στην ψηφοφορία. Οι κατοχώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, δεν ήταν και η Δανία. Νομίζω ότι και εσείς αν μη τι άλλο υπογράψατε την επιστολή ή όχι. Τέλος πάντων, σε αυτήν την επαλλαγή τρεις χώρες αποφάσισαν και ανέλησαν τι έγινε την προηγούμενη φορά που κράτησαν ε, αποχή οι χώρες αυτές και είπαν ότι τελικά το μήνυμα δεν πέρασε. Οπότε καταψηφίσαμε την απαλλαγή. Και αυτό είναι κάτι καινούριο στα πλαίσια αυτά. Λοιπόν, τι συζήτηση κάνουν από αυτού τα κράτη-μέλη, πώς αντιδρούν. Υπήρξε ένα μήνυμα που να έφτασε ε, στο Συμβούλιο και εσείς υπό την ιδιότητα της Υπουργού αλλά και υπό την ιδιότητα εκπροσώπου του Συμβουλίου. Τι έχετε να πείτε. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν η Δανία. Και έτσι θέλω να περάσω στην επόμενη ερώτησή μου. Το Ενωμένο Βασίλειο πολλές φορές είναι υπεύθυνο για σφάλματα στα προγράμματα και έχουν ένα ιδιαίτερο υψηλό ε, ποσοστό σφάλματος προσπαθούμε να συζητήσουμε κάτι που ελπίζω και εσείς να συζητάτε ή να το έχετε ήδη συζητήσει, ότι αν δηλαδή έχουμε ένα 8% λέει το λεκτικό συνέδριο ποσοστό σφάλματος και λέει ότι θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί σε επίπεδο χωρών μελών. Αν όντω είναι έτσι, τότε το Συμβούλιο τι συζητάει πάνω σε αυτό, τι λέει. Και τι λέτε εσείς στις τρεις αυτές χώρες για τις οποίες το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι είναι υπεύθυνη για το 60% περίπου του σφάλματος η Ισπανία, η Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει; Εμείς τους προσπαθήσαμε, τους καλέσαμε να έρθουν εδώ και να το συζητήσουμε μαζί τους. Δεν ήρθανε όμως. Και κάποιοι έστειλαν επιστολή και λέτε, ωραία, δεν θέλετε εσείς να έρθετε σε εμά, να έρθουμε εμεί σε εσά να το συζητήσουμε, γιατί για μα είναι σημαντικό. Τι λέει λοιπόν το Συμβούλιο, εμεί δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση στι επιστολέ που στείλαμε, ακόμα και αν ήμασταν διατεθειμένοι να ταξιδέψουμε και να πάμε εκεί. Εσεί συναντιέστε μαζί του. Και δεν είναι μόνο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποθέτω ότι είναι θέμα και των άλλων χωρών μελών. Οι άλλε χώρε μέλη πώ αντιδρούν. Το έχετε συζητήσει ε, μαζί τους το θέμα αυτό της ευθύνη των χωρών ε, μελών και ιδιαίτερα αυτών των τριών χωρών τη στιγμή που λένε ότι θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί πάρα πολλά ασφάλματα σε εθνικό επίπεδο. Και αν το έχετε συζητήσει, πού έχετε καταλήξει. Εμείς προσπαθούμε να ρωτήσουμε τους συναδέρφους σας και να μιλήσουμε. Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία, μια που είσαστε εσείς εδώ τώρα. Δράτω με τις ευκαιρίες αυτές και ρωτάω εσάς. Ελπίζω κάποιες από τις ερωτήσεις μου να μπορέσετε να μου τις απαντήσετε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε Φέλνερ. Είναι ευρύ το φάσμα των ερωτήσεων. Εγώ θα σας πρότεινα να απαντήσετε κατευθείαν σε αυτό και μετά μπορούμε να συνενώσουμε ομάδες ερωτώντων από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέλνερ για τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε εδώ. ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΙΤΗ <clears throat> εδώ σήμερα. Αλλά συζητήσαμε το θέμα αυτό σε γενικούς όρους, γιατί ουσιαστικά θέλαμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εξετάσαμε την κατάσταση κάθε κράτος πέρας για να πούμε κάνατε αυτό, δεν κάνατε εκείνο λοιπά Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι προφανώς θα ήθελα να μεταφέρω και ορισμένα από αυτά τα οποία θα προκύψουν τη συζήτηση στο Συμβουλίο ΚΟΦΗΝ για να έχουν τα μέλη του Συμβουλίου κάποια γενική εικόνα των συζητήσεων εδώ και σε σχέση με την αντίδραση στις τελευταίες συστάσεις του πρόσφατου ΕΚΟΦΗΝ. Έρχομαι τώρα στα σχόλιά σας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και την απλοποίηση. Ξέρουμε ότι όσο υπάρχουν συμβιβαστικές λύσεις σε μια πολιτική διαργασία, καταλήγουμε πάντα σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αν όλοι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν ένα πετραδάκι, τότε φυσικά έχουμε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αν έχουμε πράγματι τη φιλοσοφία και τη φιλοδοξία μιας ε, απλοποίησης σε όλες τις πολιτικές διαργασίες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι συμβαστικές λύσεις στις οποίες καταλήγουμε θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα όπως διηθούνται προς τα κάτω στο σύστημα. Το γνωρίζω αυτό και στην δανεική πραγματικότητα. Αν ζητήσετε από κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι, ίσως κάνουν και λίγο παραπάνω και θα περιπλέξουν τα πράγματα περισσότερο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ξέρουμε τι είδους φάλματα λαμβάνουν χώρα και πού η απλοποίηση θα ήταν μια καλή μέθοδος για να τα αντιμετωπίσουμε. Είπατε ότι οι τρεις χώρες έχουν καταψηφίσει. Ναι. Αλλά η προσέγγιση των τριών αυτών χωρών που αποφάσισαν να πούν όχι και να καταθέσουν μια επιφύλαξη είναι απόψεις που διατυπώθηκαν και από χώρες οι οποίες είπαν τελικά ναι λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά όλα αυτά τα θέματα και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ μιας ριζικής εκβάθρων αλλαγής και του να συνεχίσουμε σταδιακά να βασιζόμαστε στις ήδη επιτευχθήσεις ε, πρόοδους. Το δικό μου συμπέρασμα τουλάχιστον όταν εγκρίναμε αυτές τις συστάσεις ήταν ότι κάποιες από τις αντιρρήσεις των τριών χωρών, κάποιες από τις ανησυχίες των χωρών αυτό που τους οδήγησαν να καταψηφίσουν ήταν και ανησυχίες των χωρών οι οποίες υπερψήφισαν τις συστάσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα θέματα αυτά. Οι περισσότερε χώρε θεώρησαν ότι είναι πιο επικοδομητικό να συνεχίσουμε την επεξεργασία μα στη διαδικασία τη απαλλαγή και όχι με το να μην δεχόμαστε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, <clears throat> έχει δύο πλευρές το κέρμα. Κάποια πράγματα είναι θετικά, κάποια δεν είναι θετικά, κάποια προχωρούν, κάποια όχι. Δεν προχωρήσαμε σε λεπτομέρεια, λεπτομεριακή εξέταση σε όλε τι χώρε. Ήταν μια πιο γενική συζήτηση για, την, για το θέμα τη απαλλαγή. Ήταν μια καλή συζήτηση, ήταν αρκετά εκτενή και νομίζω ότι είχε ακριβώ αυτή την προσέγγιση που προσπάθησα να σα εξηγήσω. Ακολουθεί ο κύριος Ρασδάουσκας, ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά μου και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τις απαντήσεις της. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Μια πληροφορία θέλω. Συστήνει το Συμβούλιο την απαλλαγή. Άκουσα επίσης ότι συστήνει την απαλλαγή και στο ίδιο το Συμβούλιο. Οπότε ρωτάω, εσείς συστήνετε απαλλαγή στο Συμβούλιο και εφόσον ναι, βάσει ποιο εγγράφου το κάνετε αυτό. Και αν το κάνετε βάσει διαφόρων εγγράφων, θα μπορούσαμε, παρακαλώ, τα δικά σας, τα έγγραφα πάνω στα οποία βασίζεστε για να δώσετε απαλλαγή στο Συμβούλιο, τουλάχιστον αυτό συστήνεται στο Κοινοβούλιο, τα έγγραφα αυτά μπορείτε να μας τα δώσετε και εμάς. Ευχαριστούμε. Ο Φίλιπ πρώτο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη συνδρία της Επιτροπής αυτής, οπότε ε, ξέρω ότι βρίσκομαι μαζί με πιο εμπειρούς εδώ, οπότε ε, συγχωρέστε με αν δεν τα καταφέρω καλά. Ευχαριστώ πολύ πάντως την Υπουργό που ήρθε και άκουσα με ενδιαφέρον τόσα είπε. Είμαι κάπου 13 χρόνια Ευρωβουλευτής εδώ, πρώτη φορά σε αυτή την Επιτροπή πράγματι, αλλά έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια τις διαδικασίε απαλλαγή στην Ολομέλεια. Έχω την εντύπωση, η Υπουργός πολύ σωστά εντόπισε τις αδυναμίες στα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής. Από ό,τι φαίνεται όμως, έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή ακούμε ότι ναι υπάρχουν προβλήματα, ναι δουλεύουμε προσπαθώντας να τα λύσουμε, αλλά δεν λύνονται ποτέ. Και γιατί δεν λύνονται ποτέ, γιατί συνεχίζουμε να δίνουμε την απαλλαγή, οπότε φαίνεται σαν όλα να πηγαίνουν καλά. Φοβάμαι λοιπόν ότι όσον αφορά εμένα, τουλάχιστον, τουλάχιστον εκεί που εντοπίζονται περιοχές όπου το ποσοστό σφάλματος αυξάνει αντί να μειώνεται, τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να πούμε στους αυτούς μας «Ε, μήπως ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από αυτό και να προσπαθήσουμε να κοιτάμε τα ουσιαστικά ζητήματα που για μένα, και τα εντόπισε και ο κύριος Φέγιαν πριν από λίγο, εκεί όπου δεν υπάρχει πραγματικός φυσικός έλεγχος ή ελάχιστος έλεγχος, της αξιολόγησης και της δαπάνης σε προγράμματα, για παράδειγμα το Ταμείο Συνοχής ή και στην Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπέθρου, όπως είπε ο Υπουργός. Ο κύριος Φιέλεν πριν από λίγο αναφέρθηκε στο Ενωμένο Βασίλειο, τη δικιά μου τη χώρα. Μπορώ να σας πω ότι από τη δικιά μας την πλευρά, τα νούμερα έχουν να κάνουν με το 2010, η κυβέρνηση συνασπισμού προσπαθεί να τα εξετάσει, τα εξετάζει και ξέρει ότι εν μέρη οφείλονταν στον μηχανισμό που ίσχυε στον Ηνωμένο Βασίλειο και που τώρα έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί. Οπότε, επ' αυτού, αν μη τι άλλο, θα υπάρξει βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις. Πάντως, το γενικό μου σχόλιο, Πρόεδρε, όσον αφορά την παρουσία εδώ της Υπουργού, είναι ότι εξακολουθούμε να μην ε, δείχνουμε τη δύναμή μας και να μην αντιμετωπίζουμε με το στένος που θα έπρεπε τα αποτελέσματα. Εδώ θα έπρεπε να ζητάμε ε, μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή για οποιοδήποτε σφάλμα. Και όχι να λέμε δουλεύουμε για να τα λύσουμε. Όχι, το κοινοβούλιο όμως θα έπρεπε να λέει όχι, όχι και πάλι όχι, μέχρι ότου να έχουμε τα ποσοστά που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε να Ακολουθεί ο Θεόδωρος Κυλακάκης. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ θετικό που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε σε μια χρονική εποχή που όλοι θέλουν περισσότερη διαφάνεια σε όλους τους προϋπολογισμούς και ιδίως στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το ερώτημα μου είναι πολύ απλό και ως σκιώδης εισηγητής για την απαλλαγή του Συμβουλίου το θέτω αυτό υπήρξε μια επιστολή η οποία απεστάλλει από τον Πρόεδρό μας που περιελάμβανε ορισμένα ερωτήματα προς το Συμβούλιο σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής που θεωρεί για τα θέματα αυτά η νομική μας υπηρεσία ότι είναι τμήμα της γενικής απαλλαγής της Κομισιόν και αναρωτιέμαι αν το Συμβούλιο έχει την πρόθεση να απαντήσει τα ερωτήματα σε αυτή την επιστολή. Υπάρχει ήδη μια σειρά ερωτήσεων. Μπορείτε αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για το ερώτημα του κυρίου Στάς και του κυρίου Σκυλακάκη αφορούν ουσιαστικά το ίδιο θέμα πιστεύω. Και δεν έχω και την εμπειρία του κυρίου Μπράντμπερν ή την εμπειρία που θα ήθελε να έχω ο κ. Πράτμπον και εγώ είμαι νεόφερτη στα θέματα αυτά. Πάντω είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο έχει τύχει συζήτηση επανειλημμένα στο παρελθόν. Το Συμβούλιο όταν πρόκειται για την απαλλαγή αναφέρει ότι βάσει της συνθήκης το άρθρο 319 αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη βάση μιας σύστασης του Συμβουλίου θα πρέπει να δώσει <clears throat> απαλλαγή στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού, την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Ξέρω ότι υπάρχει μια διαμάχη το θέμα αυτό και δεν πρόκειται να σας απογοητεύσω λέγοντας ότι δεν θα ξεπεραστεί αυτή η διαμάχη σήμερα. Το Συμβούλιο βασίζεται για τη δική του θέση στην ε, ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν θα λυθεί όμως σήμερα το πρόβλημα αυτό της ε, διαβίβασης πληροφοριών και του ανοιχτού πνεύματος για τα θέματα αυτά. <clears throat> για το ερώτημα του αν η χορήγηση απαλλαγή είναι φραγμός στο να υπάρξει αλλαγή στα πράγματα αυτά, όταν εγώ προετοίμαζα τον εαυτό μου για <clears throat> τον ε, έλεγχο από, την, ε, το δανεικό Ελεκτικό Συνέδριο, έθεσα και εγώ αυτό το ερώτημα. Όταν υπάρχει 7,7% ποσοστό σφάλματος, αυτό είναι πραγματικά πολύ ψηλό. Όταν υποτίθεται το φράγμα πρέπει να είναι 2% το όριο. Και παρά το γεγονό ότι ο μέσος όρος σφαλμάτων είναι χαμηλότερος από το 7,7%, νομίζω είναι 4,4% μου είπαν και με πείσανε ότι αν δείτε την ε, ιστορική εξέλιξη τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Όχι ριζικά, αλλά κάθε χρόνο συνήθως κάτι γίνεται. Είτε τα πράγματα πήγαν χειρότερα και μετά πάλι καλύτερα. Συνολικά όμως υπάρχει θετική πορεία. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι στους φορολογούμενους, <clears throat> έναν το Κανείς δεν θέλει να υπάρχουν σφάλματα. Όλοι έχουμε την φιλοδοξία να αλλάξουμε το σύστημα ώστε να υπάρξει μια χωρίς επιφυλάξεις δήλωση αξιοπιστίας αλλά είναι τελικά θέμα ψυχοσύνθεσης και νοοτροπίας. Πολλοί από εμά θέλουμε να δίνουμε, να χορηγούμε την απαλλαγή και να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε αργά και συστηματικά για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Απλοποίηση, εντοπισμό, εντοπισμός των σφαλμάτων που αναδύονται ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι οι αποδέκτες των κονδυλίων θα κάνουν πιο σωστά τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος ο ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ως Θανός θα χρησιμοποιήσω την κοινή μας γνώμη, την κοινή μας γλώσσα. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, σε ποιο βαθμό το Συμβούλιο έχει συζητήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ξέρετε ότι το EFSF ε δημιουργήθηκε το 2010 και η Πορτογαλία ήταν η πρώτη η οποία επωφελήθηκε από το ταμείο αυτό και είναι αρκετά υψηλά τα, τα, τα ποσά που την χάνουν εγγυήσεων. <clears throat> Κατά τη δική μας άποψη, αυτό το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το θέμα της νομικής βάσης για τη δημιουργία του EFSF αλλά επίσης και η αξιολόγηση της λειτουργίας του και ο κοινοβουλευτικός του έλεγχος. Υπήρξαν σκέψη για τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο. Ποια είναι λοιπόν η, η θέση σας σε σχέση με αυτό το Ταμείο και τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Επανέρχομαι στο αυτό το οποίο ε, ελέγχθη. Είναι τρεις οι χώρες οι οποίες ε, απορρίπτουν την αρχή της χορήγησης της ε, απαλλαγής. Δεν είναι μία από αυτές η Δανία, ούτε και πέσει. Νομίζω ότι ήταν πριν από δύο χρόνια ή μάλλον το 2011 καλύτερα πέρσι, εμείς ως Δανία δεν είχαμε ακολουθήσει τη γραμμή η οποία εγκρίνεται φέτος. Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται είναι το εξής. Γιατί θα πρέπει εδώ να δοθεί η απαλλαγή ενώ στο παρελθόν δεν εδίδεται. Δεν εδίδεται στο σημείο αυτό. Είπατε ότι υπάρχει κάποια διαφωνία στους κόλπους των, του Συμβουλίου. Ναι, είναι τρεις χώρες οι οποίες είπαν όχι. Γιατί όμως αυτό πρέπει να μας <clears throat> οδηγήσει σε αλλαγή στις θέσεις που κράτησε στο παρελθόν το βασιλείο της Βασιλείας. Λοιπόν, είμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου τελικά φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό σφαλμάτων αντί να μειωθεί. Λέτε ναι, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι πριν από πολλά χρόνια. Βεβαίω. Αλλά κινδυνεύουμε να βρούμε του εαυτού μα σε μια κατάσταση όπου θα αυξηθεί έτσι περισσότερο το ποσοστό σφαλμάτων στο μέλλον. Και παρόλα αυτά το Συμβούλιο θα δίδει την ε, απαλλαγή ακόμα και αν τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Όλα αυτά δεν είναι κατανοήσιμα για μένα. Μου λέτε ότι προχωρούμε με μικρά βήματα. Το σέβομαι αυτό που λέτε. Αν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, μπορούμε να δώσουμε την ε, απαλλαγή. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό τη φορά γιατί αντί να υποχωρεί το ποσοστό σφαλμάτων, αυξάνεται. Τρίτο ερώτημα. Πολλές φορές η Ιδανική Προεδρία θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα διάφανη και την συγχαίρουν γι' αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτή η διαφάνεια θα μας επιτρέψει αύριο το απόγευμα όταν μιλάμε στο σημείο 46 και συζητούμε την ε, ε, απαλλαγή του Συμβουλίου αν θα είσαστε παρούσα τότε που είσαστε προσκεκλημένοι και εκεί θα τεθεί το θέμα 46 για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Σας περιμένω λοιπόν αύριο το απόγευμα κύριε Υπουργέ. Probably not. go. ahead if you like uh, with the questions. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε τώρα να αποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί θα συγκεντρώσουμε τρεις ε, ερωτήσεις. Η κυρία Γκρέσλε είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ ωραία που ήρθατε και σας ευχαριστούμε. Και μη μου θυμώσετε, αλλά έχοντας ακούσει όλα αυτά τα ωραία που είπατε, ε, αισθάνομαι σαν να είμαι εδώ ε, σε μία σάτυρα. Γιατί ξέρετε το πρόβλημα δεν υπάρχει κάπου, υπάρχει πολύ συγκεκριμένα, σε πολύ συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και υπάρχει εξής δυσάρεστη κατάσταση. Η Ισπανία εδώ και δέκα χρόνια ε, προηγείται σε όλες τις ε, αδυναμίες και ανομαλίες στα διαθροτικά ταμεία, ακολουθεί η Ιταλία και μετά η φίλη μας η Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά η διαφορά με το Συμβούλιο είναι ότι μερικές φορές εμείς το γράφουμε κιόλα. Το ερώτημα λοιπόν που δείτε είναι το εξής. Τι κάνει το Συμβούλιο για να εντοπίσει εκείνα τα κράτη τα οποία πράγματι έχουν πρόβλημα. Γιατί το θέμα δεν είναι να εντοπίσει κανεί και να σηκώσει το δάχτυλο σε συγκεκριμένου ανθρώπου και να του πει εσεί φταίτε. Το θέμα που τίθεται είναι πώ θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την ολέτρια κατάσταση όπου οι κανόνε ε, γίνονται όλο και πιο αυστηροί για όλου, ενώ κατ' ουσίαν το πρόβλημα είναι μόνο μερικοί. 2000-2006 αυτή η χρήση, η περίοδος έχει τελειώσει. Και όπως σας είπα, συνέβη αυτό που ανέφερα προηγουμένως και ο Επίτροπος μας το επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία και πάλι είναι πρωταθλητής. Ε, τώρα βέβαια προηγείται η Ελλάδα και νομίζω μετά ακολουθεί η Τσεχία. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε ένα πρόβλημα πάντα με τα ίδια κράτη-μέλη. Κάποια στιγμή λοιπόν οφείλουμε να λάβουμε ειδικά μέτρα για αυτά τα κρατημέλη και γι' αυτό ερωτώ. Προβλέπονται ειδικά μέτρα για τα κράτη που εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος επανειλημμένα στα διευθυντικά ταμεία, δηλαδή ειδικά μέτρα για Ισπανία και Ιταλία. Τώρα, όσον αφορά τα τελευταία κράτη που προσεχώρησαν, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που αναμφίβολα βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Βλέποντας λοιπόν την τελευταία έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και πρόσφατη μάλιστα. Στη Ρουμανία έχουμε την εξής κατάσταση. Διαφθορά 60%. 60% των περιπτώσεων που αφορούν διαφθορά αναστέλλονται. Σε τελική ανάλυση, τι γίνεται, σε ορισμένα κράτη δείχνουμε κάποια ανοχή, αλλά η διαφθορά ισχύει παντού, υπάρχει παντού. Δεύτερον, στη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 27 ποινικέ διαδικασίες κατά ε, ενός μεγάλου αριθμού δικαστών. Ε, και στην Γερμανία υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς στην Δανία, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχουμε λοιπόν δύο κράτη-μέλη με φοβερά προβλήματα και ρωτώ, τι ακριβώς ε, κάνει το Συμβούλιο όσον αφορά στη διαχείριση των κονδυλίων, ειδικά όσον αφορά αυτά τα θέματα, ποιο είναι το σχέδιο που υπάρχει. Και θα ήθελα να πω και το εξή η ε, απόφαση απαλλαγής με εντυπωσίασε πάρα πολύ, διότι η απόφαση αυτή περιλαμβάνει και ορισμένε ε, σημαντικές ε, προτάσεις. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ειδική έκθεση για τις ανακτήσεις στη γεωργική πολιτική, στην οποία εργάστηκα και εγώ. Αυτή η ειδική έκθεση είναι 8 γραμμές. Σε κάποιες άλλες ειδικές εκθέσεις ε, έχουμε 2-3 σελίδες, αυτό δεν το βρίσκω σωστό. Βέβαια, σε αυτές τις 8 ε, γραμμές ε, καθίσατε σαφές ότι το πρόβλημα και πάλι αφορά συγκεκριμένα κράτη-μέλη, τα οποία δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που έχουν αναλάβει με βάση το κοινοτικό δίκτυο, δίκαιο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που μπορώ να το πω και σε πολύ λίγα λόγια ότι αυτό είναι το θέμα. Ε, τι είδους προγράμματα έχετε για να βελτιώσετε το σύστημα ανακτήσεων. Νομίζω ότι ε, πρέπει και εσείς εργαστεί με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Κατανοώ ότι αυτό είναι δύσκολο για εσάς, αλλά ξέρετε αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ε, το, αυτό απαιτεί η συγκεκριμένη ε, στιγμή, δηλαδή να μην προσποιούμε ότι όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα, να θέσουμε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλε. Επόμενος είναι άλφος κύριος Γκάια. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό. Δεν είναι πολύ συχνά που έχουμε αυτή την χαρά και την τιμή να έχουμε υψηλού επίπεδο εκπροσώπους του Συμβουλίου στην Επιτροπή μας χαιρόμαστε για το θέμα αυτό, αλλά βλέπετε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν <clears throat> πολλά σχόλια από την Επιτροπή μας που δείχνουν την ε, ματέωση που νιώθουν πολλά μέλη της Επιτροπής μας. Για το γεγονός επίσης ότι εμείς ως κοινοβουλευτικοί και ιδίως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ δεν έχω ερώτημα, έχω περισσότερο ένα σχόλιο. Θα Είναι σχόλιο αυτό το οποίο ήθελα να σας αναφέρω και θα ήθελα να έχω την άποψή σας σχετικά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο μέσα σε ένα συμβούλιο που έχουμε 27 κράτη να είναι τα 26 κράτη παραγωγός χάρη ειλικρινή με ένα, άλλο, με ένα κράτος το οποίο έχει προβλήματα στην, ε, προϋπο, στην ε, Έχουμε όλοι προβλήματα οικονομικά αυτή τη στιγμή και να πρόκειται στο Συμβούλιο να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν διορθωτικές πορείες στα κράτη αυτά, ώστε να μπορέσουμε όλοι να λειτουργήσουμε καλά σε μια ε, ένωση και σε μια οικονομική, σε μια ευρωζώνη επίσης. Πρέπει όμως το σύστημα αυτό να μην το οποίο ακολουθείται από το Συμβούλιο να μην οδηγεί σε ανευθυνότητα σε ορισμένα κράτη. Γιατί πολλές φορές δίδονται ε, απαλλαγές για κράτη-μέλη τα οποία έχουν μια αντιμετώπιση η οποία δεν ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν θέματα βέβαια τα οποία πρέπει να επιληφθεί το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ καταρχήν για τα κράτη-μέλη, αλλά παραμένουν και τα ζητήματα που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε για περιπτώσεις που γίνονται σφάλματα ή ατασταλίες έναντι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά ο φορολογούμενος ο Ευρωπαίος πληρώνει για σφάλματα άλλων και όχι για σφάλματα στα οποία οι ίδιοι οι εκπροσωποί του υπεύθυνοι. Ένα από τα βασικά θέματα είναι τα θέματα των διαθωτικών πόρων, των, ε, ε, του Περιφερειακού Ταμείου ιδιαίτερα, που είναι η αχίλιος πτέρνα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για μένα, η περιφερειακή πολιτική βρίσκεται σε επιμερισμένη διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη έχουν να συμμετάσχουν στη διαχείριση και επομένως τα σφάλματα προέρχονται κυρίως και από τα κράτη-μέλη. Και όταν έρχονται τα θέματα αυτά στο ΕΚΟΦΗΝ, τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνω μια τελείως διαφορετική στάση και να μην δεχτούν αυτά τα σφάλματα τα οποία έχουν διαπράξει. Κύριε Μπράτμπορ, λοιπόν, πρέπει εσείς να πάτε στην κυβέρνησή σας και να πείτε ότι και η δική, η δική σας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία από τη μια μεριά θέλει να υπάρξει έλεγχο των σφαλμάτων, από την άλλη μεριά συμμετέχει ιδιαίτερα στα σφάλματα αυτά, στην διάπραξη των σφαλμάτων. Για μένα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει το εξή, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα σφάλματα που βρίσκονται στην επιμερισμένη διαχείριση. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα, μέσα που έχει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εάν δούμε ότι το, τα σφάλματα δεν πέφτουν κάτω από το 2% ή κοντά στο 2%, θα πρέπει να ζητήσουμε στην Κομισιόν, στο Κοινωνικό Ταμείο και αντίστοιχα στο Περιφερειακό Ταμείο να τους παροτρύνουμε να διακόπτουν τα προγράμματα στα οποία παρατηρούνται τέτοιου επίπεδου σφάλματα. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την Κομισιόν να προχωρήσει σε αναστολή ή σε διακοπή προγραμμάτων που είναι υπερβολικό, υπερβολικά ψηλό το ποσοστό των σφαλμάτων για να επιτευθεί η προστασία των φορολογουμένων. Αυτή είναι μία δυνατότητα. Και Η, η άλλη δυνατότητα είναι να υπάρξει και η ανάκτηση αυτών των ποσών που δίδονται από την Κομισιόν. Ναι. Θα πρέπει να μειώσουμε τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν ε, στα κράτη-μέλη ουσιαστικά με την ε, σιωπηρή αποδοχή του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να παραγνώσουμε το γεγονός ότι υπεύθυνο για την ε, μείωση των σφαλμάτων στα κράτη-μέλη είναι το ίδιο το Συμβούλιο. Τα κράτη λοιπόν τα οποία ψήφισαν κατά της απαλλαγής κατά κάποιο τρόπο έχουν καταψηφίσει τον ίδιο τον εαυτό τους. Και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα βρούμε ένα κοινό τρόπο με όλα τα κράτη-μέλη για να μειώσουμε το ποσοστό των σφαλμάτων. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τρεις πολύ σοβαρές ερωτήσεις αυτές που αντικατοπίζουν τις συζητήσεις που έχουμε στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω. Αυτό μου θύμισε την ταινία Καζαπλάκα, Ingrid Bergman και Humphrey Bogart. Στο τέλος λέει... Να, η απάλληλη είναι ύποπτη. Ίσως μπορείτε πάντως να απαντήσετε σε αυτές τις σοβαρές ερωτήσεις που ακούστηκαν. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι στο τέλος ίσως να λέει επίσης ότι μπορεί να είναι η αρχή μιας πολύ όμορφης φιλίας. Και ίσως θα έπρεπε έτσι να το δούμε. Γιατί όταν προετοιμάστηκα για την συνάντηση αυτή, Είχα στο μυαλό μου διάφορα πράγματα μπορεί κανείς να πει για το ποσοστό σφάλματος. Μπορεί να πει κανείς σε μερικούς τομείς είναι υψηλότερο φέτος, σε άλλες είναι όπως θα έπρεπε να είναι, που δείχνει δηλαδή κάποια πρόοδο για να πάμε προς το επιθυμητό 2%. Και μπορούμε βέβαια να προχωρήσουμε και να βρούμε μια χρονιά που να δείχνει ότι τα πράγματα είναι πιο καλά από ό,τι κάποια άλλη. Και να χρησιμοποιήσουμε αυτή σαν σημείο αναφοράς και σύγκρισης. Για μένα πάντως πρέπει να δούμε ποια είναι η διαδικασία που θα μας κατευθύνει στο σωστό σημείο. Στο Συμβούλιο δεν βλέπουμε να έχει νόημα το να καταδεικνύουμε κάθε φορά τον ε, υπεύθυνο naming and shaming. Υπάρχουν δυσκολίες τεχνικές, διοικητικές και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάνει ό,τι μπορεί να κάνει επ' αυτού. Γι' αυτό και τα πράγματα αλλάζουν. Σε μερικές περιπτώσεις. Αυτό που λέει η κυρία Γκρέσλερ φυσικά και είναι πολύ σωστά. Ότι δηλαδή οι ανακτήσεις από δημοσιονομικές διορθώσεις είναι κάτι πολύ ουσιαστικό για να μπορούμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ κεντρικό πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες για τις ανακτήσεις από διοσυνομικές διορθώσεις, για να γίνονται οι διορθώσεις αυτές. Οι κανόνες και οι μηχανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά γιατί τότε θα μειωθούν και τα ποσοστά ασφάλματος. Το έχουμε δει αυτό μέχρι τώρα και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και στο μέλλον. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Προφανώς κάθε βουλευτής, υπουργός, πρόεδρος, οποιαδήποτε επιτροπή εννοείται ότι θέλει να μπορεί να κοιτάει τους ε, Ευρωπαίους πολίτες στα μάτια και όχι να τους δείχνει ότι δεν τον νοιάζει. Πολύ σημαντικό αυτό. Συγχρόνως, η άλλη πλευρά της συζήτησης είναι να δούμε πώς θα αποφύγουμε τα προβλήματα. Να μην προκύπτουν δηλαδή, να καταπολεμούνται στην ρίζα τους. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε αυστηρά μια πολιτική διακοπής, παύσης, πληρωμών ευθύς εξ αρχής. Κάθε φορά δηλαδή που διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία. Και να μην γίνονται πληρωμές μέχρι να υπάρξει διόρθωση. Και είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο λέει πως υπάρχει περιθώριο για παρετέρω βελτιώσεις και στους δύο τομείς και πρέπει να γίνουν. Το τονίζει ιδιαίτερα για να έχουμε ε, αξιόπιστη ενημέρωση όσον αφορά τις ανακτήσεις από τις νομικές ε, διορθώσεις που γίνονται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το ξέρουμε αυτό ότι υπάρχει δρόμος που συστήνεται εδώ και αυτόν πρέπει να πάρουμε. Βέβαια μπορεί κανείς να ρωτηθεί ναι αλλά πώς μήπως δεν πρέπει να συστήσουμε την απαλλαγή λένε κάποιοι. Εγώ όμως πώς βλέπω τα πράγματα. Βελτιώνονται. Και νομίζω ότι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουμε και επικεντρωμένοι στην απλοποίηση και στην τεχνική αρρωγή, να συνεχίσουμε και έτσι θα έχουμε συνεχή βελτίωση. Αυτό χρειαζόμαστε, βελτίωση χρειαζόμαστε. Έτσι θα την έχουμε. Συνεπώς, είμαστε σε κάποιο σημείο που πρέπει να διαπιστώσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να επικεντρωνόμαστε εκεί που πρέπει να υπάρξει παρετέρω βελτίωση. Θέλω να πω κάτι άλλο για το EFSF, τον προσωρινό μηχανισμό δηλαδή κρίσης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν μπαίνει σε αυτά τα πλαίσια. Θα εξεταστεί περιμένουμε τον μόνιμο μηχανισμό που θα αρχίσει από το καλοκαίρι, γιατί η συνθήκη ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μόνο όσον αφορά τον μόνιμο μηχανισμό. Κάτι το οποίο αφήνει περιθώρια για συζήτηση. Όπως είπα και νωρίτερα σε μια άλλη ερώτηση, δεν νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα κοινοβούλιο-συμβόλιο σε αυτήν τη συνεδρίαση. Δεν πιστεύω και το νομίζω ότι θέλει κανένα από εμά να ξαναφτιάξουμε τη συνθήκη από την αρχή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Τσέσκοβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο εδώ και να ρωτήσω μερικά πράγματα και να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την προβληματική αυτή που εξετάζουμε. Βλέπετε, έχω την αίσθηση ότι στη συνεδρίαση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ότι κατά κάποιο τρόπο βγάζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα στορό στολίδια και αρχίζουμε με το καθένα να ασχολούμαστε. Όμω, εγώ δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Αναφερθήκατε στην. Μια συνάδελφο αναφέρθηκε στη Τσεχία και είπε ότι υπάρχουν οι αμαρτωλοί μεταξύ άλλων και η χώρα μου λοιπόν. Αλλά εγώ κάποια στιγμή στην Ολομέλεια πήρα το λόγο και είπα ότι η τσεχική δημοκρατία αναφέρεται στην ετήσια αυτή έκθεση, για πρώτη φορά αν δεν απατώμε, για κάποιες αδυναμίες που εντοπίστηκαν. Και θα ήθελα να ακουστεί ξεκάθαρα το τι συμβαίνει και όσον αφορά τα αποτελέσματα της διαχείρισης, αλλά και όσον αφορά τα σφάλματα στη διαχείριση και την εφαρμογή των ε, κανόνων που διέπουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια διότι έχουμε και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και με κάθε σεβασμό που αξίζουν η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, γιατί εγώ πάω διακοπές σε αυτές τις χώρες πολύ ευχαρίστω. συχνά. Ερεύνησα λίγο τα πράγματα, μελέτησα Και από ό,τι φαίνεται, το ποσοστό σφάλματος και άλλα θέματα τα οποία αναφέρονται εδώ, σχετικά με την Τσεχία, ε, λοιπόν αυτά δεν ε, δικαιολογούν να αναφέρεται η Τσεχία. Στην συζήτηση αυτή λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις χώρες εκείνες οι οποίες αποτελούν μέρος της Ευρωζώνης και από την άλλη μεριά να δούμε τις χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, έχουν το δικό τους εθνικό νόμισμα. Έχω λοιπόν μία ερώτηση. Γιατί στην Επιτροπή μας εδώ πρόσφατα συζητήσαμε σε τι βαθμό μπορούμε να στηρίξουμε το ρόλο της ε, τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και είπαμε στην Επιτροπή μας εδώ ότι τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να στηριχθούν από όλες τις χώρες μέλη. και να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τα διαφορετικά ταμεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις χώρες μέλη. Και γιατί, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα βοηθήσει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όπως ονομάζεται, και κινδυνεύει να χάσει τα τριάλφα της. Θέλω λοιπόν να ξέρω ποιες είναι οι εξελίξεις, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα για το μέλλον. Γιατί βλέπετε υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που τις έχω ακούσει και που δεν ξέρω αν παίζουν εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τσέσκοβα. Και <clears throat> λόγω του ότι περνάει η ώρα, ε, προτείνω να περάσουμε στον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων και καταρχής, ε, καταρχήν μία παρατήρηση επιτρέψτε μου όσον αφορά αυτό που αναφέρθηκε για τους αμαρτωλούς. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια θρησκευτική έννοια και πρόσφατα διάβασα ότι όλοι οι Άγιοι έχουν παρελθόν και όλοι οι αμαρτωλοί μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε και από καθαρά θεολογική σκοπιά, ε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Γιατί το θέμα δεν είναι να επιτεθούμε σε ορισμένους, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιτύχουμε βελτίωση. Να το επιτύχουμε από κοινού. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Είναι βέβαια σημαντικό ε, το να επισημάνει κανεί ε, τους υπεύθυνου ε, για να προβούν και αυτοί σε απαραίτητες βελτιώσεις. Εμείς ως κοινοβούλιο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όπως σας είπα να θέσουμε το δάκτυλο στον τύπο των ήλων. ε, άλλους δύο έχω νομίζω, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον και αν όχι θα ήθελα ε, να κλείσω τον κατάλογο των ερωτών σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Δεν πήρα απάντηση στην ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ. Ειλικρινά μιλώντας, είναι γελίο να μην βρίσκεται εδώ το Συμβούλιο. Ακούσαμε πολλές θέσεις από το Συμβούλιο. Έχουμε εκπροσώπους του Συμβουλίου που ήρθαν μετά τη συζήτηση. Δεν φαίνεται να βελτιώνεται η σχέση Κοινοβουλίου-Συμβουλίου. Μπορεί το Συμβούλιο να μην έχει να πει πολλά πράγματα. Μπορεί το Συμβούλιο αύριο να έρθει να μας πει ναι, αλλά υπάρχει συνθήκη. Κατά την ταπεινή μου γνώμη όμως, το καλύτερο θα ήταν να έρθει το Συμβούλιο εδώ, αύριο το απόγευμα. Και ένας λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα δεν ήθελε να δώσει απαλλαγή στο Συμβούλιο είναι γιατί διαπιστώνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή κακή θέληση. Δεν υπάρχει καλή θέληση από πλευρά του Συμβουλίου να προχωρήσει σε διάλογο μαζί μας. Έπειτα, κανείς δεν θέτει σε αμφισβήτηση ε, το γεγονός ε, ότι το Κοινοβούλιο δίνει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Η απαλλαγή αυτή πρέπει να δοθεί επειδή δίνουμε απαλλαγή στην Κομισιόν. Τότε δίνουμε στην Κομισιόν απαλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να τη δώσουμε υποχρεωτικά και στο Συμβούλιο. Μαζί πάνε αυτά. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ένα μέρος του προπολογισμού του Συμβουλίου καλύπτεται από την Κομισιόν. Ναι, αλλά εξής ποιο ρωτάτε. Την Κομισιόν ή το Συμβούλιο. Αν ρωτήσουμε την Κομισιόν, είναι περίπλοκα τα πράγματα. Είναι προτιμότερο να μπορούμε να μιλήσουμε κατευθείαν με το Συμβούλιο. Και εκεί είναι που γίνονται, που μπερδεύεται το πράγμα. Γιατί κανονικά, κανονικά, ε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια εξαίρεση. Η Σουηδική Προεδρία ήταν μια εξαίρεση, γιατί εκείνη θέλησε να μιλήσει μαζί μας και το έκανε, άρα είναι εφικτό. Η Σουηδική Προεδρία μας έδωσε γραπτά απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Τις, βάλαμε στην ιστοσελίδα, τις στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Δηλαδή μπόρεσε το Συμβούλιο να απάντησε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλει, μπορεί το Συμβούλιο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα άλλο. Τώρα, πέρα από την ε, Προεδρία του Συμβουλίου, δεν καταφέρνουμε να έχουμε και εξηγήσει για τα πιο στοιχειώδη ζητήματα. Και μια ερώτηση που συστηματικά τίθεται κάθε χρόνο είναι πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο να βάζει παραπάνω χρήματα στον προπολογισμό του για την μετάφραση, για παράδειγμα. Πάντα στη μετάφραση μπαίνουν παραπάνω χρήματα στον προπολογισμό του Συμβουλίου. Και όχι μόνο αυτό, κάθε χρόνο ζητούν και αύξηση του προπολογισμού για τη μετάφραση, παρόλο που δεν έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα κονδύλια τα οποία είχαν δοθεί την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει, συμφωνώ να είναι ένα αποθεματικό για την πολιτική για τα κτίρια, ναι, αλλά γιατί. Γιατί. Εδώ δεν βλέπουμε τα ποσά για την μετάφραση. Εμείς θέλουμε τα ποσά. Μήπως θα μπορούσε ο υπουργό να μας τα δώσει. Με είναι εκνευριστικό, γιατί πρόκειται για εκατομμύρια ευρώ. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Τι θέλετε, εγώ τι, πώς θέλετε όλα αυτά να τα πουλήσω στους εκλογείς μου και να τους πω ότι είναι εντάξει λογαριασμοί. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Με πληροφόρησαν μόλις ότι η κυρία Υπουργός θα πρέπει να φύγει στις 4 και 4 για να προλάβει το αεροπλάνο της. Κύριε Φιέλνερ, αν μπορείτε να είστε πάρα πολύ σύντομος. Είπατε στην αρχή ότι θα μεταφέρετε τα διαμυφθέντα στη συζήτηση αυτή πάλι στο Συμβούλιο. Αυτό είναι μια ευκαιρία για μας. Και είπατε επίσης ότι δεν περνάτε από τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ πρέπει να περάσετε μέσα από τα κρατη αυτό είναι το μήνυμά μας. Όχι για να τους επωνυδίσετε και να τους καταδείξετε ποιοι είναι οι, αυτοί οι οποίοι έχουν, κάνει, έχουν δημιουργήσει τα σφάλματα, αλλά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο γιατί τα περισσότερα σφάλματα πράγματι προχωρούν, προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Και δεν μπορείτε να το επιλύσετε το πρόβλημα αυτό αν δεν προχωρήσετε σε πιο έντονες ενέργειες. Μια επιμερισμένη διαχείριση σημαίνει επιμερισμένη ευθύνη και όχι αποποίηση ευθύνης. Και όπως λέει και η κυρία Γκρέσλε, χρειάζεται ένα πραγματικό σύστημα ανάκτησης <clears throat> και όταν προσαρμόσετε το νέο πρόγραμμα για το Ταμείο Συνοχής, ελπίζουμε ότι εσείς θα μπορέσετε να τονίσετε αυτά τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι είσαστε ικανοί στις κυρώσεις και στα θέματα ε, Μην αφήσετε λοιπόν μονάχα του Υπουργού Ανάπτυξη να μιλάνε για αυτά τα προβλήματα στην επόμενη περίοδο σχεδιασμού. Χρησιμοποιήστε την εμπειρία σα και μεταφέρετε τα στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέλλερ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αύριο το Συμβούλιο θα εκπροσωπείται, όχι από μένα βέβαια. θα υπάρχει κάποιος υψηλό αξιωματούχος της Δανικής Προεδρίας για να εκπροσωπεί το Συμβούλιο. Και ίσως τα σχόλια τα οποία έχουν διατυπωθεί θα πρέπει να είναι ενάψιμο για την αναζήτηση λύσεων. Γιατί όταν γίνονται συζητήσεις οι οποίες είναι δύσκολες συζητήσεις και όταν ξέρουμε όλοι ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν ένα παλιό ιστορικό, ίσως θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε να έχουμε διάλογο, θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαία συμφωνία. Αυτό είναι το νόημα του διαλόγου, <clears throat> να υπάρχει και μια κοινή συνένεση. Και κάτι τέτοιο χρειάζεται όταν Πρόκειται για τη συζήτηση για το πώς θα ερμηνεύσουμε τη διατύπωση των συνδικών. Να βρούμε μια κοινή συμφωνία για τα θέματα αυτά. Και δεν νομίζω ότι μια τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σε μια αίθουσα όπως αυτή. Και επίσης για το θέμα της ε, δακτυλο... του να δακτυλοδείξουμε και να επωνυδίσουμε εαυτούς και αλλήλους, εγώ έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Η δική μου εμπειρία είναι ότι για να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να δώσετε στους ανθρώπους την ευκαιρία την υποστήριξη, τις συμβουλές για να αντιμετωπίσουν επικοδομητικά αυτά τα οποία δεν λειτουργούν, αντί να τους πείτε ότι είσαστε αμαρτωλοί ή ότι θα πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που κάνετε. Πρέπει να επιτύχουμε ένα κοινό στόχο και πρέπει να βρούμε τρόπους να επιτύχουμε όλο αυτό το κοινό στόχο. Αυτό σε ό,τι αφορά τις, ε, τις ε, διορθώσεις σε σχέση με τα δημοσιονομικά σφάλματα. Για, το, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από ό,τι ξέρω το ελεκτικό συνέδριο δεν έκανε καθόλου σημειώσει για το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχει συζητηθεί αλλού η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να προωθήσει σχέδια και προγράμματα στι χώρε όπου λειτουργεί. Μπορεί να ασφάλω αλλά αν σας δώσω μια αυθόρμητη αξιολόγηση της κατάστασης, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να συμβάλλουμε περισσότερα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί η υψηλή αξιολόγηση, το τριπλό α της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με κάθε τρόπο γιατί είναι πολύ σημαντικό για το επιχειρηματικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων. Επειδή ξέρω ότι ορισμένοι αρχηγοί κρατών ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλλει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης και ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι τα σχόλια της κυρίας Τσέσκοβα για την τσεχική δημοκρατία είναι αξιοσημείωτα γιατί δείχνουν σαφώς ότι μπορούν να βρεθούν πιο επικοδομητικοί τρόποι από το να αλληλοεγκαλούμεθα και να λέμε ότι κάποιοι είναι αμαρτωλοί και κακοί και κάποιοι όχι. Για το Συμβούλιο τώρα και για τη δυνατότητα του Συμβουλίου. Να συντάξει σωστούς προϋπολογισμούς. Από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο έχει ήδη για το 2012 έχει ξεκινήσει προσπάθειες <clears throat> να μειωθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια στις γραμμές του προϋπολογισμού, ώστε να ανταποκρίνονται και να ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές ανάγκες. Θα σταματήσω εδώ. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον εισηγητή. Πράγματι, θα κάνω αυτό που είπα στην αρχή. Θα μεταφέρω όλα αυτά που είπατε στο Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και το Συμβούλιο να ξέρει πώς αντιμετωπιστήκαν οι συστάσεις του Συμβουλίου από το Κοινοβούλιο. Και επίσης, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι τα μέλη του Συμβουλίου συμμερίζονται πλήρως την αντιμετώπιση μας ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα μειωθούν τα σφάλματα και θα έχουν μονάχα ε, ίσονα χαρακτήρα και σε αριθμό και σε επίπτωση. Εξ ονόματος όλης της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βεστάγκερ για την παρουσία σας. Την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Και ίσως είναι μια η αρχή, η απαρχή μιας θαυμάσιας φιλίας που θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και χρηστή χρησιμοποίηση των δημοσίων κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, wir können. Um, if we like uh, here on this topic, uh, we can please. Um, I would like to invite uh, Commissioner Shemeta, if you. Να ζητήσω από τον Επίτροπο κύριο Σέμετα, εάν θέλει να κάνει κάποια σχόλια για το τμήμα αυτό της διαδικασίας απαλλαγής. Πρωτού, μπει στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Υπουργό για την πολύ καλή της ομιλία και θα ήθελα σε γενικές γραμμές επίσης να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία της Δανίας ε, για τα συμπεράσματα τα οποία εξήγε από αυτή τη σύσταση που καταθέτει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο καλωσορίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών. Και επίσης αναγνωρίζει ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες, ε, κυρίως σε τομείς που είναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις. Τώρα, ε, ποικίλει η εικόνα ε, στους διάφορους τομείς της ε, πολιτικής. Σε ορισμένους τομείς μπορέσαμε να σταθεροποιήσουμε τα καλά αποτελέσματα. Σε άλλους τομείς, κυρίως στον τομέα της σύνοχης, το 2010 αναχαιτίστηκε η θετική πορεία και σήμερα οι περισσότερες συζητήσεις επικεντρώνονται στην πολιτική σύνοχης και επίσης και στις ευθύνες που έχουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ε, τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους σε ε, τομείς επιμερισμένης διαχείρισης. Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στη βελτίωση και λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ε, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Κομισιόν λυπάται που τρία κράτη-μέλη δεν γκρίνουν την απαλλαγή. Παρ' αυτά, ορισμένες από τις ανησυχίες τους όσον αφορά την έλλειψη απόδοσης ορισμένων κρατών μελών και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν έγκαιρα στοιχεία από εθνικές αρχές. Επίσης, ε, θεωρεί η Κομισιόν ότι η κατάσταση ε, θα βελτιωθεί στο μέλλον με τις προτάσεις της και έτσι ε, θα καταστεί δυνατόν και τα κράτη αυτά να προσχωρήσουν στη μεγάλη πλειοψηφία που εγκρίνει τη σύσταση του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλιστεί η εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές ε, της ε, χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Και αυτό μπορεί να γίνει βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και απλουστεύοντας αυτές όπως ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δημοσιονομικό κανονισμό και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βράχει πρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει ε, να εξετάζει τις αδυναμίες που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του ελληνικτικού Συνεδρίου αλλά και στη σύσταση επαλλαγής του Συμβουλίου. Η επόμενη κρίσιμη φάση για περαιτέρω βελτίωση μακροπρόθεσμα είναι η έγκριση ε, του δημοσιονομικού κανονισμού και της ε, ε, διαρθρωτικής ε, νομοθετικής βάσης για το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Η Κομισιόν καταθέτει πολύ φιλόδοξες προτάσεις για την καλύτερη χρήση των κοινωτικών κονδυλίων και για τον εξορθολογισμό διορθωτικών μηχανισμών. Το, η σύσταση απαλλαγής του Συμβουλίου αναφέρει πολλούς τομείς όπου είναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις και συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένη προσέγγιση την οποία θα αμελητή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έτσι τελειώσαμε με το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 5. Παρακαλώ. Α, κύριε Κρέσλερ, για το 4 ακόμα. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία του Επιτρόπου για να σας μεταφέρω μια είδηση. Εχθές σε μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με το πακετό για την Όλαφ. Καταλήξαμε σε ένα έγγραφο. Έτσι ελπίζω το κείμενο αυτό ε, να το στείλουμε σήμερα το βράδυ στους συντονιστές. Εν πάση περιπτώσει ε, θα έχουμε όλες τις θέσεις και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση της Όλαφ. Και ήθελα να σας το πω αυτό σαν είδηση γιατί είναι μια καλή είδηση ε, που θεωρώ ότι τη θέλετε κι εσείς γιατί σας είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κρέσλε, λέει ο πρόεδρος, ε, κατόπιν τούτου. Κλείνουμε το σημείο υπαριθμών 4 της μέσης διάταξης. Πάμε στο 5, είναι πάλι στο ίδιο θέμα. Ε, και σας ερωτώ ε, κατά πόσο ενδεχομένω στο σημείο αυτό ε, θέλετε να πείτε κάτι για το σημείο υπαριθμών 5 ή μήπως πρέπει να δώσουμε το λόγο απευθείας στον εισηγητή. Θα έλεγα το λόγο, καλύτερα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Φιαλίνα και μετά θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, είμαι πάντα έτοιμος. Πρώτα απ' όλα, έγραψα την έκθεσή μου Εντάξει, δεν ε, έχω τελειώσει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το κύριο κομμάτι της δουλειάς ε, για μένα έχει γίνει. Βρίσκεται πίσω μου. Μας μένει δουλειά να κάνουμε, δεν λέω. Λοιπόν, υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή πρώτα απ' όλα για να σας ευχαριστήσω όλους. Να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και τις υπηρεσίες του Ελεκτικού Συνεδρίου. Με βοήθησαν πάρα πολύ ε, ακόμα και σε απίθανες ώρες τους έπαιρνα τηλέφωνο για να τους ζητάω σημειώματα για το ε, χύψη. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντούν στις ερωτήσεις μου επικοδομητικά. Οι πληροφορίες δηλαδή που μου έδωσαν, πάνω στις οποίες βασίστηκα, ήταν πολύτιμες. Ευχαριστώ επίσης και τον Μπεν και τον Χριστόφ της Γραμματείας Χωρίς αυτούς δεν θα είχα μπορέσει να ετοιμάσω την εκθεσή μου. Ο βοηθός μου ψιθυρίζει, μου λέει μην ξεχάσεις να πεις ευχαριστώ και για μένα, ε. οπότε ναι, ευχαριστώ και αυτόν. Όντως, είχα κοντέψει να τον ξεχάσω. Αυτός δεν είναι ο λόγος που έχει κανείς ε, βοηθούς για να σου θυμίζουν πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ λοιπόν και εσένα. Λοιπόν, απόφαση για την απαλλαγή. Υπάρχει κάτι καλό. Για την απόφαση της απαλλαγής πρέπει να σας πω ότι μου τηλεφώνησε κάποιος ο οποίος είχε διαβάσει την έκθεση και μου είπε εντάξει όλα τα καταλάβαμε αλλά υπάρχουν τρεις τελίτσες που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνουν αυτές οι τρεις τελίτσες? Μα ακριβώς. Πολύ σωστό το ερώτημα. Ακριβώς. Παραμένει ανοιχτό το Άννα θα αντιδώσουμε την απαλλαγή ή αν θα την αναβάλουμε. Και γιατί, γιατί η ετήσια έκθεση του λεκτικού συνεδρίου διαπιστώνει αδυναμίες στην διαχείριση από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η δικιά μου η προσέγγιση και που την έχω συζητήσει και με του σκιώδες εισηγητές, οπότε δεν θα του εκπλήξει, όταν είδαν την έκθεση τουλάχιστον, στην παράγραφο 1 θα δείτε ότι αναφέρονται δράσεις προτεραιότητας για την Επιτροπή και στην ε, πρόταση για απαλλαγή αυτή θα εξαρτηθεί από τις τέσσερις δράσεις. Από αυτό και από τη φιλοδοξία που θα δείξει η Επιτροπή για αυτές τις δράσεις θα εξαρτηθεί η απαλλαγή. Οπότε εγώ λέω τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα απαλλαγή σε αυτό το στάδιο και θα επανέλθουμε. Ίσως όμως θα ήταν καλό να δει κανείς αυτές τις δράσεις προτερότητας και να τις εξετάσει κάπως. Η πρώτη δράση προτεραιότητας είναι στην παράγραφο 19. Πρόκειται για ένα θέμα που έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και είναι η χρησιμοποίηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνική αυτή, το ξέρουν οι συνάδελφοι. Εμείς πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει αρκετή ενημέρωση όσον αφορά για την χρησιμοποίηση των μέσων αυτών χρηματοοικονομικής τεχνικής. Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής θα κληθούν να παίξουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνεπώς, η καταπροτεραιότητα δράση είναι πληροφορίες να έχει ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, αξιολόγηση της πληροφορίας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να δούμε τι μαθήματα θα πάρουμε για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και τέλος, ε, να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η χρηματοοικονομική αυτή τεχνική που είναι μέσων υψηλού κινδύνου, όπως λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι χτες όλα τα μέλη της Επιτροπής μας πήρε ένα έγγραφο από την Επιτροπή ακριβώς για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και χαίρομαι γι' αυτό. Θα το μελετήσω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είχα το χρόνο, αλλά έτσι με μια πρώτη ματιά που έριξα διαπίστωσα ότι ο στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει στη διάθεσή του την πληροφορία και είναι πολύ καλό γιατί ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου όταν ετοίμασα και τη διατύπωση αυτή εδώ. Θα μας βοηθήσει λοιπόν, άρα κάτι από αυτά που ζητάμε φαίνεται να το παίρνουμε. Είναι καλό λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακούσαμε και πριν, θέλει να ενισχύσει τους κανόνες και την εφαρμογή ε, των ρυθμίσεων για την χρήση των μέσων αυτών στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Βλέπετε όμως το τρέχον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Μερικέ φορές έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή λειτουργεί βάσει δοκιμών και λάθους. Ότι δηλαδή η θεωρία των μέσων αυτών είναι πιο σημαντική από την εφαρμογή τους. Εγώ θα ήθελα αντί να η Επιτροπή να δουλεύει βάσει του δοκιμή και λάθος, να δουλέψει βάσει των πληροφοριών που έχουμε για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έτσι ώστε να προλάβει σφάλματα στο μέλλον. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ευκαιρία να δουλεύει χρησιμοποιώντας καλύτερες πληροφορίες και ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και φαντάζομαι ότι με τις πληροφορίες που θα υπάρχουν περισσότερο θα γίνει αυτό. Δεύτερη προτεραιότητα που είχε να κάνει με την παράγραφο 34. Πρόκειται για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ε, αλυσίδας λογοδοσίας. Και εδώ το Ολεκτικό Συνέδριο έχει εντοπίσει ελλείψεις και αδυναμίες της ετήσιας εκθέσεις. Η άποψη του εσωτερικού ελέγχου τη Κομισιόν επικρίθη από, την, ε, από το Ελληνικό Συνέδριο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο, μεγάλο περιθώριο βελτίωση σχετικά με την λογοδοσία στην ε, διαχείριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτή τη δράση λοιπόν εγώ περιμένω, δεν ξέρω και οι υπόλοιποι φαντάζομαι, μια πολιτική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να δέχεται την ευθύνη όσον αφορά την εφαρμογή του προπολογισμού και να υπογράφουν οι επίτροποι της της δραστηριότητες. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Και νωρίτερα το κοινοβούλιο μας ζήτησε από τους επιτρόπους να υπογράφουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Ακούσαμε ότι η επιτροπή θέλει η Γενικός Διευθυντής να το κάνει αυτό και όχι επίτροπη. Και πέρυσι πετύχαμε κάποια βελτίωση. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να υπογράψει και αν μη τι άλλο να λέω ότι το έχει συζητήσει με τους επιτρόπους του. Ε, καιρός είναι να υπογράψει και ο Επίτροπος και να λέει «Ναι, και εγώ άκουσα αυτά που μου είπε ο Γενικός Γραμματέας». Αυτό θα ήταν το επόμενο βήμα. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ως δράσεις προτεραιότητες είναι ότι οι αιτήσιοι λογαριασμοί γίνονται βάση αντικειμενικότητας και αποφεύγοντας ε, υπεραισιόδοξες ε, εκτιμήσεις. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες της ε, Κομισιόν για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το ποσοστό σφάλματος. Ζητάω επίσης να έχουμε και την γνωμοδότηση του εσωτερικού ελεγκτή. Και τέλος, θέλω να δω πώς, τι κάνει για τον ιδιωτικό τομέα επιτροπή. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρουμε ότι δουλεύει ε, για το τι κάνουν οι κυβερνήσεις με τα κονδύλια που παίρνουν, αλλά θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε και κάτι από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και η, Επιτροπή έχει να μάθει από αυτά. Και θα μπορούσε, ενδεχομένω δεν ξέρω, θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω πώς θα αποδειχθεί με το σφάλμα, θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ή όχι. Τρίτη δράση προτεραιότητας έχει να κάνει με την αυξημένη χρήση της προχρηματοδότησης. Αυτά θα τα δείτε στην παράγραφο 46. Το ελεγκτικό συνέδριο εντόπισε δύο θέματα σχετικά με την προχρηματοδότηση. Πρώτα απ' όλα ότι έχει αυξηθεί πολύ από το 2005 μέχρι το 2010 και δεύτερον ότι η προχρηματοδότηση έχει επιπτώσει στο ποσοστό σφάλματος. Ιδιαίτερα στην πολιτική εξωτερικής ε, βοήθειας. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο κίνδυνοι από την αύξηση αυτή της προχρηματοδότησης. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει υψηλότερο κίνδυνο στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος ε, δεν ε, μπορεί να πληρώσει, είναι φερέγγιος, και δεύτερον ότι μπορεί να υπάρξει αναβολή για μια ημερομηνία αργότερα που σημαίνει ότι τα σφάλματα δεν μπορούν να αποφευθούν ή να εντοπιστούν έγκαιρα εφόσον υπάρξει αναβολή για αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω δύο δράσεις προτεραιότητας. Πρώτον, ενημέρωση του Κοινοβουλίου, γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση στη χρήση της προχρηματοδότησης, ήταν ένα μόνιμο ερώτημα που είχαμε μετά από την πρώτη φορά που συζητήσαμε με τους συναδέρφους σας για τομείς όπου είχαμε διαπιστώσει αύξηση της προχρηματοδότησης. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι η προχρηματοδότηση θα πρέπει να μειωθεί μόνο στο απόλυτα αναγκαίο επίπεδο. Για νέα δηλαδή προγράμματα. Τέταρτη δράση προτεραιότητας είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κυρώσεων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό το έχουμε συζητήσει και με την Υπουργό, το συζητήσαμε μάλλον στο προηγούμενο σημείο μας. Το έχουμε συζητήσει και με τον Επίτροπο Χάν. Εκτενώς. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο ελέγχει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Εξακολουθώ να έχω και εδώ δύο ερωτήσεις. παρά τη συζήτηση. Το πρώτο είναι, έχει μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, εάν ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει χρησιμοποιήσει. Σε αυτό το στάδιο προσπαθώ να απαντήσω σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και καταλήγω στα Πρώτον, κάποια μέσα δεν είναι αποτελεσματικά ή τουλάχιστον όχι αρκετά αποτελεσματικά. Αυτό ισχύει νομίζω για τις περισσότερες δημοσιονομικές διορθώσεις που τι γίνεται, οι χώρες αντικαθεστούν κάποια προγράμματα με άλλα προγράμματα, οπότε τελικά αυτή η δημοσιονομική διόρθωση είναι εικονική, δεν γίνεται πραγματικά. Άλλα πάλι μέσα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Δηλαδή δεν προχωράει σε διακοπή ε, των κονδυλίων. Και αυτό το βλέπουμε ότι παρά τις όποιες διακοπές έχουν γίνει, το ποσοστό σφάλματος αυξάνει. Και γνωρίζουμε σήμερα ότι η Επιτροπή γνωρίζει πού ε, εντοπίζονται τα περισσότερα σφάλματα. Μένω δηλαδή με την αίσθηση ότι οι πληρωμές γίνονται ίσως υπερβολικά γρήγορα σε σχέση με το τι ξέρουμε για τα σφάλματα και που θα μπορούσαμε να κάνουμε διακοπή της χρηματοδότησης. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι μένα με ξέπληξε που δεν είχε υπάρξει διακοπή για το 2010 για το Ταμείο Συνεχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου ξέρουμε ότι υπήρξε αύξηση του σφάλματος. Κατέληξα λοιπόν όταν πρόκειται για τις δράσεις προτεραιότητας και τις ε, κυρώσεις το εξή. Ότι η Επιτροπή ίσως θα έπρεπε να υποστηρίξει αυτά που λέει το Κοινοβούλιο για έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου και κυρώσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο τουλάχιστον. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης επιλέξιμων προγραμμάτων από νέα προγράμματα. Ακόμα και αν αυτά είναι επιλέξιμα. Τουλάχιστον να γίνεται πολύ λιγότερο από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα η αντικατάσταση αυτή. Και δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να προχωρούν στην ανάκτηση των ποσών από τους δικαιούχους για να μην αναγκάζονται να πληρώνουν δύο φορές. Τα είχαμε πει αυτά και στα πλαίσια της έκθεσης Χατζημαρκάκη. Τώρα οι κανόνες για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την πολιτική συνοχής, αποδοτικά και οικονομικά. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται ιδίως σε περιοχές οι οποίες επανειλημμένα έχει αποδειχθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Αυτό είναι το μάθημα που παίρνουμε, ότι επαναλαμβανόμενα παρουσιάζονται προγράμματα στις ίδιες χώρες, μερικές φορές ακόμα και στην ίδια περιφέρεια της ίδιας χώρας και μάλιστα και στα πλαίσια των ίδιων προγραμμάτων σε αυτές τις περιφέρειες. Τώρα η αναφορά των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ασκεί ε, το δικαίωμα ελέγχου που έχει καλύτερα. Αυτά είναι τα σημεία που είχα να σας δείξω όσον αφορά τις δράσεις προτεραιότητας για την Επιτροπή. Τώρα μπορεί να υπάρξουν και τροπολογίες και από μένα ως εισηγητής. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει ε, την έκθεση εξολόγησής τη στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Το περιμέναμε. περιμέναμε και περιμέναμε αυτή την έκθεση εξολόγησης. Και έτσι σαν πρώτο πράγμα πρέπει να σας πω ότι δεν έχω εντυπωσιαστεί. Παρ' όλα αυτά είναι καλό. Είναι δύσκολο να πούμε «Α, επιτέλους πήραμε την αξιολόγηση» επιβεβαιώνει πάντως 20 Μαρτίου θα έχουμε συζήτηση, δηλαδή πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Λέει όμως στη συνθήκη ότι πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Οπότε, λέω, δεν είναι δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό εμείς καλά τη στιγμή που για πρώτη φορά θα συζητήσουμε την αξιολόγηση αυτή στις 20 Μαρτίου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Θα προσπαθήσω πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα να τα καταφέρω με την εξέταση αυτή της πρώτης εκδοχής της έκθεσης αξιολόγηση. Είναι και η πρώτη φορά, οπότε, οπότε θα γίνει. Τέλος, τέλος, τέλος. Θέλω να υπενθυμίσω ότι θα έχω κάποιες τροπολογίες για αυτά τα οποία συζητήσαμε και με την Υπουργό. Όπως είπα και πριν, και ε, η κυρία Γκέριν και ο κύριος Χατζημαρκάκης, μετά βέβαια ανέλαβε ο κύριος Μέλντερ ως σκιώδης από το Άλτε, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν το ταξίδι απαλλαγή, όπω το ονομάσαμε, για να δούμε πώ ε, μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση των δαπανών. Επίσημα λοιπόν ζητήσαμε να έχουμε κάποιες επαφές και επίσημα δεν πήραμε καμία, απόφαση, καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Νομίζω ότι ο Βρετανός Υπουργός τι έκανε. Έστειλε. Α, μα ζήτησε να του ξαναστείλουμε ξανά και ξανά το ίδιο πέντε φορές γιατί κάθε φορά έλεγε ότι το έχανε. Τη Μαγιόρκα, Πορτοφίνο και Μπράιτον. Χτες πάντως αποφασίσαμε να μην κάνουμε τότε που είχαμε υπολογίσει να το κάνουμε αυτό το ταξίδι γιατί δεν προλαβαίναμε έτσι καλλιώς. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα το θέμα αυτό θα το θέσουμε. Τη συμμετοχή δηλαδή των κρατών μελών. Και θα επανέλθουμε σε αυτήν την ιδέα να πάμε εμείς και να έρθουμε σε επαφή στις χώρες αυτές που πρέπει με τους αρμόδιους. Θα επανέλθω λοιπόν με τροπολογισμούς σε αυτά τα δύο σημεία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περιμένω τα δικά σας σχόλια. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ο Χριστόφορος Φέλνερ είναι ο εισηγητής και μου είχε ζητήσει η γραμματεία καθώς προχωράει με σε διάταξη να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις και να προχωράμε στα επόμενα σημεία να συζητήσουμε καταρχήν το 5 και 6 από κοινού όπως βλέπετε είναι αλληλένδετα δεν ξέρω αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις μπορούμε να συζητήσουμε το 5 και το 6 μαζί δεν βλέπω καμία αντίρρηση Και δίνω και το λόγο στον κύριο Σεμέτα για μια πρώτη απάντηση. Έχετε το λόγο κύριε Σεμέτα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Φέλνερ για το σχέδιο εκθεσής του. Ήδη από την αρχή της διαδικασίας απαλλαγής υπήρξε μια πολύ επικοδομητική ε, προσέγγιση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και η Κομισιόν ήταν πάντα έτοιμη να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τις ε, πρώτες μας ε, αντιδράσεις στις περιοχές προτεραιότητας που εντοπίζει ο εισηγητής σας στο σχέδιο έκθεση. Η πρώτη δράση προτεραιότητας αφορά την εφαρμογή και τον έλεγχο των εργαλείων χρηματοπιστωτικής μηχανικής, όπως λέγεται, που χρησιμοποιούνται για τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό το οποίο μας αφορά καταρχήν ως πέριμνα είναι η αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου αυτών των εργαλείων που γίνεται μέσω ε, εποπτείας και λογιστικού ελέγχου. Μπορώ σας πω με χαρά ότι το ρινό ρυθμιστικό πλαίσιο θα ενισχυθεί ιδιαίτερα με τις τροπολογίες στον αντίστοιχο κανονισμό που εγκρίθηκαν το προηγούμενο δεκέμβριο από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη τώρα έχουν υποχρέωση τακτικής παροχής ε, εκθέσεων σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά αυτά εργαλεία. Η Κομισιόν θα αρχίσει από τα μέσα του 2012 να παίρνει συγκεκριμένα στοιχεία από τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Το νέο αυτό μέσο θα περιλαμβάνει ένα, μια περιγραφή των ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων και των τρόπων εφαρμογής, την ε, ταυτοποίηση των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται, το επίπεδο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και τα ποσά αρρωγής που δίδονται στους τελικούς αποδέκτες. Επί τη βάση αυτών των στοιχείων η Κομισιόν θα συντάξει την πρώτη ετήσια έκθεση για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία τον Οκτώβριο του 2012. Επιπλέον υπήρξε ένα σημείωμα κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2011 που διευκρινίζει τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα στα κρατη σε σχέση με την αργία τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία από το 2007. Πήρατε και μια επιστολή χθε από τον Ιωάννη Χάν και εμένα τον ίδιο, που περιλαμβάνει μια πλήρη ανάλυση αυτών των χρηματοπιστωτικών εργαλείων, τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει και τα μέτρα που έχει λάβει η Κομισιό στην τωρινή προγραμματική περίοδο για τη βελτίωση αυτών των εργαλείων και για το μέλλον επέκεινα αυτή. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο η Κομισιόν προτείνει να έχει ενισχυμένους μηχανισμούς παρακολούθησης αυτών των εργαλείων και χαιρετίζει και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι η διαδικασία η δομή ευκυβερνησίας μέσα στην Κομισιόν. Το θέμα αυτό συζητήθηκε ήδη στην διαδικασία απαλλαγή του 2009. Έκτοτε έχουν έλθει σημαντικέ βελτιώσει στον τομέα αυτό, ιδίω σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του συστήματο εποπτεία και διαχείριση τη Κομισιόν. <clears throat> Τον ε, περασμένο Νοέμβριο υπήρξε και μεταρρύθμιση των μονίμων εντολών σε σχέση με την εκπόνηση αυτή τη έκθεση και καλύπτει τα περισσότερα από τα στοιχεία που έδειξε ο εισηγητή. ιδίω δόθηκε πρόσθετη, <clears throat> δόθηκαν πρόσθετες κατευθύνσεις σε σχέση με την εκτίμηση του υπολοιπόμενου επίπεδου σφαλμάτων και των δυνητικών κινδύνων. Στις πρόσφατες συζητήσεις μας, μετά από τις συζητήσεις αυτές, το σχέδιο ε, έκθεση απαλλαγής ζητάτε να αναφέρονται και τα συμπεράσματα της Κομισιόν στην έκθεση αυτή. Το σύστημα <clears throat> λογοδοσίας που έχουμε βασίζει τη διαδικασία αξιοπιστίας σε ένα σαφή διαγωνισμό μεταξύ του πολιτικού επίπεδου και του διαχειριστικού επίπεδου. Αυτή η δομή διακυβέρνησης δεν έχει διαφυσβητηθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Αντίθετα, η Κομισιόν αναγνωρίζει την ανάγκη να καταδείξει ότι αυτή η ίδια ως συλλογικό σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων που στη συνέχεια εκχωρείται η ευθύνη στους γενικούς διευθυντές και στις υπηρεσίες τους. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, η Επίτροπη έχει ζητηθεί να συναντώνται τακτικά με τους γενικούς διευθυντές τους, τουλάχιστον δύο ειδικέ συναντήσεις στον χρόνο, να συζητούν τα θέματα λογιστικού ελέγχου, ατασταλιών και ε, απατών και να εξετάζουν και την ετήσια έκθεση. Επίσης, οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει να επικυρώνουν επίσημα στην έκθεσή τους, στην ετήσια έκθεσή τους, ότι τα κύρια στοιχεία αυτής της έκθεσης και η δήλωση αξιοπιστίας μαζί με την οποία όλες οι ε, ενστάσεις και επιφυλάξεις έχουν συζητηθεί με τον αρμόδιο επίτροπο. Και επίσης όλες οι δηλώσεις των γενικών διευθυντών θα πρέπει να περιέχουν και μια σαφή δήλωση προς την κατεύθυνση αυτή. Λαμβάνουμε υπόψη επίσης το γεγονός ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει την πλήρη πολιτική ευθύνη για το έργο των Γενικών Διευθυντών και Υπηρεσιών επί τη βάση των δηλώσεων και επιφυλάξεων που διατυπώνται στην ετήσια έκθεση. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να εγκρίνεται σε μία από τις εβδομαδίες συναντήσεις της Κομισιόν μετά από την πλήρη ε, εξέτασή της από τους Επιτρόπους. Η Κομισιόν θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο αυτή την άσκηση λογοδοσίας και θα εξετάσει οποιασδήποτε προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, ο Γενικός Ελεκτής της Κομισιόν προσκλήθη πέρσι από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου για να εξετάσει δυνητικές αλλαγές που θα προσθέταν αξία στην όλη αυτή η διαδικασία και έτσι θα αντανακλούσαν καλύτερα την επαγγελματικότητα και την ανεξαρτησία του όσοι υπεύθυνο για το λογιστικό έλεγχο στο εσωτερικό της Κομισιόν. Έρχομαι τώρα στα θέματα προχρηματοδότησης που αναφέρθηκαν στην τρίτη, στην τρίτη προτεραιότητα δράσης. Η αύξηση προχρηματοδότησης δικαιολογείται από τις ανάγκες καταβολής κονδυλίων στη νέα αυτή περίοδο προγραμματισμού και την επιμερισμένη διαδικασία διαχείρισης. Η Κομισιόν θα πληροφορήσει εν περισσότερο, εν περισσότερο λεπτομέρεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δράσεις προχρηματοδότησης από το 2005 έως το 2010 η Κομισιόν συμμερίζεται την άποψη ότι η προχρηματοδότηση χρειάζεται να έχει μια ειδική προσοχή. Πρέπει να βρεθεί μια συμβαστική λύση η οποία εξασφαλίζει ότι θα πάρουν τα απαραίτητα χρήματα οι αποδέκτες για να υπάρξει η εκκίνηση των προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως προστατεύονται τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρέπον επίπεδο προχρηματοδότησης λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες ε, χρηματοδότησης και τους εμπλεκόμενους κινδύνους και την ε, διάρκεια των προγραμμάτων και τα μέτρα τα οποία υπάρχουν για τον έλεγχο των θεμάτων αυτών. Η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και έχει προτείνει ένα επίπεδο προχρηματοδότησης στο νέο κανονισμό. Στην συνάντηση του Ιανουαρίου 2012 βρέθηκε μια συμβαστική λύση η οποία προβλέπει τώρα μια προσέγγιση κόστους ωφελίας σε σχέση με την τακτικότητα της διαδικασίας ε, συμψηφισμού για τις ε, προχρηματοδοτήσεις και ένα σύστημα το οποίο καλύπτει χωριστά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η τέταρτη δράση προτεραιότητα ζητά τη δημιουργία ενό αποτελεσματικού μηχανισμού κυρώσεω στον τομέα τη πολιτική συνοχή. Συμφωνεί η Κομισιόν ότι τα εργαλεία για την παρακολούθηση τη εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχει εντοπίσει στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη δράση της Κομισιόν σχετικά. Να αναφέρω μονάχα τις κύριες αλλαγές οι οποίες προτείνονται από την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, η εισαγωγή δημοσιονομικών διορθώσεων προς τα κράτη-μέλη εάν υπάρξουν σημαντικές ε, ατασταλίες οι οποίες διαπιστώνονται από την Κομισιόν ή από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δεύτερον, συνθήκες και προϋποθέσεις κάτω από τις μπορούν να ανασταλούν ή να διακοπούν οι πληρωμές. Επίσης, οι διακοπές μπορούν να ισχύουν για 9 μήνες και όχι 6 μήνες όπως τώρα και θα είναι πιο αναλογικές προς το αντίστοιχο τμήμα των πληρωμών που καλύπτουν τα προβλήματα. Επίσης, η αντιμετώπιση των φορέων που θα πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μέσα στα πλαίσια των προγράμματων. Η Κομισιόν προτείνει ορισμένα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν την πρόληψη των σφαλμάτων και θα ευθυγραμμίσουν καλύτερα τους μηχανισμούς για τα κονδύλια αυτά, όπως είναι η ετήσια δήλωση αξιοπιστίας και η πιστοποίηση των αντιστοίχων φορέων σε εθνικό επίπεδο και επίσης μια, περισσότερη, μια μεγαλύτερη χρήση του λεγόμενου απλοποιημένου κόστους η πρόταση αυτή σαφώς αποκλεί τη δυνατότητα των αρχών διαχείρισης να επιλέγουν προγράμματα πριν να γίνει η ε, απόφαση χρηματοδότησης τα λεγόμενα αναδρομικά προγράμματα. Επίσης αντιμετωπίζονται τα, τα προβλήματα εκθέσεων στα κράτη-μέλη. Προληπτικά, η μελλοντική διαδικασία ελέγχου στην Κομισιόν για το επίπεδο εκτέλεσης των προγραμμάτων θα περιλαμβάνει και μια έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές καθυστερήσεις ή αναδυόμενα προβλήματα. Η Κομισιόν όμως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει επικοδομητικά οποιασδήποτε προτάσει ή ιδέες στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το νέο δημοσιονομικό, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα μπορούσαν να βελτιώσουν με καλή σχέση κόστου κόστος-οφέλεια στην διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι τώρα στην ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που αφορά τα πορίσματα και τις συστάσεις. Η έκθεση του Κοινοβουλίου αφορά αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτό το νέο στοιχείο της διαδικασίας απαλλαγής που εμφανίζεται για δεύτερη φορά είναι πράγματι πάρα πολύ εύστοιχο. Το ελεκτικό συνέδριο έκανε ελέγχους για θέματα διαχείρισης και αυτά ήταν σημαντικά στοιχεία που μας βοηθούν να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την ε, επίδοση στα συστήματα της Κομισιόν. Αυτοί οι έλεγχοι μας βοηθούν να εντοπίσουμε πού βρίσκονται αδυναμίες στη σχεδίαση των συστημάτων ή στην εφαρμογή τους και ποιες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα, με ένα τρόπο που είναι εποφελής σε σχέση με το κόστος ώστε να μειωθεί το επίπεδο σφαλμάτων και να μην έχουμε επιφυλάξει σε σχέση με την τελική δήλωση. Η Κομισιόν θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά όλα αυτά τα οποία ζητά το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ειδική αυτή έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, έντιμα μέλη, η Κομισιόν είναι πάντα έτοιμη να υπομειστεί τις ευθύνες της σε σχέση με την εκτέλεση του προεπολογισμού. Σας έχω παρουσιάσει ένα σχέδιο, ένα αδρό διάγραμμα του πώς βλέπει η Κομισιόν το μελλοντικό της έργο για να αντιμετωπίσει τις εντοπιζόμενες αδυναμίες και να επιτύχει τις προσδοκόμενες βελτιώσεις. Στο επόμενο διάστημα, σε επόμενες μέρες, θα επιβεβαιώσω και εγγράφος τη δέσμευση της Κομισιόν στα κύρια αυτά σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και θα το πράξουμε πιο λεπτομεριακό τρόπο. Εν κατακλείδη θέλω να υπογραμμίσω την πλήρη προσήλωση της Κομισιόν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα, όλες τις δράσεις ε, προτεραιότητες που αναφέρονται στο ψήφισμα περί απαλλαγής. Ευχαριστούμε κύριε Σεμέτα. Τρεις θέλουν να λάβουν το λόγο συνάδελφοι. Ο κύριος Γκάιερ είναι πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή δουλειά που έκανε και που ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον κοινό μας ε, στόχο που είναι να ε, περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος ε, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μας είπε περιλαμβάνουν πάρα πολλές καλές ιδέες. Έχει και τέσσερις πολύ καλές προτεραιότητες και τον ευχαριστώ βέβαια και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τους ε, συντονιστές. Αυτοί εντάχθηκαν πάρα πολύ καλά ε, σε όλη τη διαδικασία και πολύ συχνά συζητήσαμε για το τι θα συμπεριλάβουμε από την έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη, πώς αυτά θα τα εξελίξει περαιτέρω ο κύριος Φέλγνερ και πώς ε, θα ενταχθούν όλα αυτά ε, στη ε, σύσταση για απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προέκυψε μια θαυμάσια συναδελφική σχέση που ελπίζω να συνεχιστεί επί της ουσίας και στο μέλλον. Κατόπιν τούτου, όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Φέλνερ, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω να κάνω ουσιαστικές παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι όπου εμείς ως πολιτική ομάδα έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη. Γιατί αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το είχαμε ήδη πει στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Βεβαίως και ε, εγώ θα καταθέσω τροπολογίες γιατί υπάρχουν κάποια σημεία στη διατύπωση που πρέπει να ομολογήσω ότι μας φαίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά. Ε, στο τέλος, ας πούμε, προς το τέλος της έκθεσης υπάρχει ένα σημείο όπου λόγω των ε, δυσκολιών ε, που υπάρχουν ε, στους κανισμούς κρατικών προμηθειών είναι δύσκολο να λειτουργήσει η κοινή αγορά και αυτό δεν θέλουμε να το στηρίξουμε. Κατά τα άλλα, επιτρέψτε μου να αναφέρω τέσσερις προτεραιότητες. Θα είμαι σύντομος και σαφής είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις τέσσερις προτεραιότητες. Εμείς ε, στηρίζουμε τις ε, προτάσεις του κυρίου Φέλνερ για τα χρηματοδοτικά μέσα. Στηρίζουμε στο σύνολό τους αυτές τις προτάσεις. Διαβάζοντας όμως τις προτάσεις αυτές, μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα που θα πρέπει λιγάκι να το δούμε, δηλαδή πώς μπορούμε να εφεύρουμε έναν τέτοιο μηχανισμό έτσι ώστε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία όταν ακολουθούν λάθος κατεύθυνση να μπορούμε να τα αναστείλουμε. Η υποχρέωση ενημέρωσης είναι σωστή, όμως μπορούμε να φανταστούμε να υπάρχει και ένα είδος φρένου. Δεν ξέρω τώρα πολιτικά πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ίσως ε, πρέπει να εξοικειωθούμε περισσότερο με τα θέματα και αυτό προτιθέμεθα να το κάνουμε ως ε, Επιτροπή. Αλλά αυτό προέκυψε και από τη συζήτηση που μόλις είχαμε για το ποσοστό σφάλματος ε, στον τομέα της ε, συνοχής. Αλλά λοιπόν ε, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να πει τώρα αναστέλουμε, διακόπτουμε και εμείς να μπορούμε ως Κοινοβούλιο να υποβάλουμε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει μία διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό το είδος φρένου εισαγωγικά θα πρέπει να υπάρχει στα χρηματοδοτικά εργαλεία σε τελική ανάλυση σε άλλα θέματα αν αυτά βοηθούν ε, εμείς συμφωνούμε αλλά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό, αυτά αναφέρεται στη συνθήκη και αναφέρεται και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο να κάνει αυτή τη δήλωση. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι και η Κομισιόν το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα στι προχρηματοδοτήσει, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο προβληματικά. Γιατί επενεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον ε, στα περιφερειακά ταμεία. Αυτό βέβαια δεν είναι το επίκεντρο των εργασιών του συνομιλητή, αλλά ε, κατεβλήθησαν προσπάθειες ε, με, από κοινού με τον εισηγητή να αντιμετωπιστεί κάποια ύφεση, κάποια μείωση, γιατί αυτό είναι και δικό μας καθήκον ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός ε, όσον αφορά τις ε, προχρηματοδοτήσεις. Δεν θα ε, αμφισβητούσα με τέτοια σαφήνεια όπως το πράττει ο κύριος Φέλνερ τις προχρηματοδοτήσεις. Βεβαίω και δεν πρέπει να υπάρχει ποσοστό κινδύνου, επ' αυτού συμφωνούμε απόλυτα, αλλά θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Να δούμε λιγάκι και τις πολιτικές προεκτάσεις των προχρηματοδοτήσεων. Και όλα αυτά να μην τα καταδικάζουμε συλλήβδιν. Και κάτι άλλο, ένα δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Συζητάμε τώρα με το Συμβούλιο έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ε, ανάγκης ε, να επανέλθει το θέμα της ε, επιμερισμένης διαχείρισης γιατί αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο πρόσφατα. Ασχοληθήκαμε μια ολοκληρή μέρα με το εν λόγω άρθρο. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το Κοινοβούλιο ε, έδωσαν μάχη κατά του Συμβουλίου όπου θελήσαμε ε, να πείσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου ο οποίος ε, δεν αισθανόταν στο τέλος ε, και πολύ άνετα, αλλά δεν είχε εντολή από το Συμβούλιο να υπερασπιστεί αυτό το θέμα της επιμερισμένης διαχείρισης. Αν λοιπόν είχαμε μία μελέτη η οποία θα προήρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταδείκνυε το πώς ακριβώς μπορούμε να περιορίσουμε το ποσοστό λάθους στην πολιτική συνοχής, αν δηλαδή αποκλίνουμε από τις προχρηματοδοτήσεις. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα είχαμε και ένα μέσο πίεσης προς το Συμβούλιο, όπου θα μπορούσαμε να τους πούμε, κοιτάξτε, ανεξάρτητοι ελεγκτές ή αν θέλετε οι εμπειρογνώμες κομισιών καταλήγουν ε, στην εξής αξιολόγηση κινδύνου. Και λόγω αυτού, αυτό θα ήταν το επόμενο πολιτικό βήμα, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς για να αναχαιτίζουμε προχρηματοδοτήσεις έτσι ώστε να περιορίζουμε τους ε, κινδύνους. Θα πρέπει να στηρίζουμε την ε, ε, ανάπτυξη. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για το θέμα του κινδύνου που συνδέεται με τις προχρηματοδοτήσεις. Και εάν τελικά αυτό είναι ένα μέσο πίεσης απέναντι στο Συμβούλιο, ε, αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, συστήνω τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται τα ποσοστά λάθους ήδη στα κράτη-μέλη, το να αντικατασταθεί αυτό το σύστημα, αυτό ε, σας προειδοποιώ, ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλά λάθη, σφάλματα μάλλον, θα μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί ήδη ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην μιλάμε για οργανωμένη ανευθυνότητα. Στη τελική ανάλυση όλοι επιθυμούμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Όμω, αφού το θέλουμε αυτό, θα πρέπει πρέπει να πούμε ότι οι δυνατότητες που έχει το κράτος μέλος, οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν. Ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος και το επόμενο ε, πρόγραμμα ε, να είναι λανθασμένο, αλλά εγώ είμαι υπέρ της αρχής ε, ότι ισχύει αθότητα μέχρι αποδείξεως ε, του εναντίου. Τώρα, αν πρόκειται για προγράμματα του παρελθόντος, εκεί πράγματι είμαι υπέρ της, ε, του διεξοδικού ελέγχου. Γιατί συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πάρα πολλά, εδώ θίγονται πάρα πολλά θέματα, όπως και το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης ε, αξίας. Εγώ λοιπόν λέω το εξής ότι αν δεν καταφέρουμε να το πράξουμε αυτό σε αυτή την έκθεση, να το πράξουμε στην επόμενη. Να δούμε λοιπόν ε, ποια ε, λάθη μπορούν να υπάρχουν σε παρελθόντε προγράμματα και να εξετάσουμε προσεκτικά αυτά αλλά ε, τη δυνατότητα μεταφοράς ε, κονδυλίων μέσα ε, στο κράτος, στο κράτος μέλος, αυτή τη δυνατότητα θέλω να την διατηρήσουμε, γιατί αν καταργηθεί θεωρώ ότι κάτι θα ήταν λάθος. Επόμενος συνάδελφος, κύριος Μούλντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε σε, μια, σε ένα ετήσιο ετήσια άσκηση που κάνουμε κάθε χρόνο και η οποία βέβαια μας φορτίζει με την δήλωση αξιοπιστίας και την απαλλαγή και έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα στον κόσμο είναι όλο και πιο δύσκολο κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο να εξηγεί γιατί δίνει την απαλλαγή. Την τελευταία φορά που δεν τη δώσαμε οι συνέπειες ήταν ε, τρομερές. Δεν θα έπρεπε όμως αν φέτος δεν δώσει απαλλαγή να υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παρατεθεί η Επιτροπή. Πάντως, διαπιστώνουμε κάθε χρόνο ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, όχι όμως αρκετή για να δώσει θετική δήλωση αξιοπιστία στο ελεγκτικό συνέδριο. Και αυτό είναι πρόβλημα για το Κοινοβούλιο. Και έχει δίκιο ο εισηγητής που το αφήνει ανοιχτό το τι θα κάνουμε, γιατί και στη δικιά μου πολιτική ομάδα πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε τι θα ήταν το καλύτερο να κάνουμε. Δεν ξέρουμε. Πολλοί βέβαια δεν θέλουν να αρνηθούμε την απαλλαγή, αλλά ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Τώρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Μία από τις συνέπειες όταν δεν δώσαμε απαλλαγή τελευταία φορά ήταν ότι δηλώθηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις δαπάνες. Και αυτό είναι στην καρδιά του προβλήματος. Και γι' αυτό ακριβώς στη συμφωνία του 2006 υπάρχει τα συμφωνία με τα κράτη-μέλη ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει ετησίως να κάνουν δήλωση με την οποία να λένε ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για την χρηστή ε, διαχείριση των κονδυλίων. Μόνο τέσσερις χώρες όμως το κάνουν τώρα και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να επαναλαμβάνει το αίτημά του και το κάνει ότι κάποιος πρέπει να έχει την πολιτική ευθύνη στα κράτη-μέλη και να κάνει τη δήλωση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει, λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει δήλωση που δίνουν ε, τα κράτη-μέλη, που ονομάζεται Annual Summary, το Φεβρουάριο κάθε χρονιάς, οπότε το κράτος μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη που του ζητάμε. Ναι, αλλά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρόβλημα είναι ότι που είναι αρχή της απαλλαγής, είναι ότι οι δηλώσεις αυτές είναι απόρριτες. Μία λοιπόν από τις τροπολογίες της ομάδας των φιλελεύθερων θα είναι να μην είναι απόρριτες οι δηλώσεις αυτές. Γιατί δεν είναι απόρριτες δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου δεν είναι απόρριτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει κανένα απόρριτο, οπότε γιατί να ισχύει αυτό. Άρα θέλουμε διαφήνεια, σαφήνεια και τέλος κάτι άλλο που απασχολεί πάντα τους φιλελεύθερους είναι ότι όταν τα ζητάμε αυτά από τα κράτη-μέλη να ξέρετε ότι τα ζητάμε και από την Επιτροπή. Ο Επίτροπος είπε ότι από πλευρά της Επιτροπής μία συνθετική έκθεση ε, μπορεί να γίνει συλλογικά να λαμβάνει την ευθύνη έτσι καλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ όμως δεν βλέπω για ποιο λόγο ένας γενικός ε, να υπογράφει κάτι το οποίο δεν δέχεται να υπογράψει συλλογικά το Σώμα των Επιτρόπων. Δεν βλέπω γιατί. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό ένας ε, γενικός γραμματέας και να μην μπορεί να το κάνει το Σώμα των Επιτρόπων. Είναι πολιτική ευθύνη. αλλά και αυτό πρέπει να το συζητήσω ακόμα στην ομάδα μου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει κάποιες εγγύησεις, χωρίς όμως να ξέρει κανείς ποιος είναι υπεύθυνο. Υπάρχει το θέμα των 60 εκατομμυρίων στον μηχανισμό σταθερότητας που θα μεταφερθούν στο μόνιμο μηχανισμό από 1η ε, Ιουλίου. Πότε είναι. 1η Ιουλίου, έτσι, ναι. Πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πρόκειται για 60 δις. Το μισό του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Ρωτήσαμε την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την δυνατότητα ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να είναι πολύ αισιόδοξη η άποψη της νομικής υπηρεσίας γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν στο ESM τα χρήματα αυτά είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ θέλω έλεγχο όχι μόνο για τα 60 δισεκατομμύρια, αλλά και για τις εγγύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς κλπ. κλπ. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς εγγυόμεθα κάτι ως κοινοβούλιο στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, ενώ κάθε φορά που πρόκειται για εφαρμογή, για χρήση, δεν μπορούμε ούτε να την ελέγξουμε, ούτε να αντιδράσουμε σε αυτήν. Γι' αυτό το σημείο λοιπόν θέλω τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 20 δισεκατομμύρια δίνονται σε εγγύησεις από τη λέω και ας υποθέσουμε ότι κάτι πάει στραβά. Μία από τις χώρες μέλη πτωχεύσει τα 60 δισεκατομμύρια, τι γίνονται. Πώς θα δαπαθούν τα χρήματα. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γι' αυτό. Είναι μια πιθανότητα κι αυτή και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Και αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες διαδικασίες που έχουμε, με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, δεν ξέρουμε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα είναι εντάξει, αλλά για μας αυτό είναι το κέριο ζήτημα. Στον προπολογισμό αυτό και στη δημοσιονομική ε, διαδικασία φέτος, αυτά είναι που μας απασχολούν και είναι και κάτι άλλο το οποίο με εκπλήσει, πρέπει να το πω και αυτό είναι θετικό. Τα μεγάλα προβλήματα όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο, ιδίως το Κοινωνικό Ταμείο. Τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου διαπιστώνουμε ότι δαπανούνται πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει το ίδιο ποσοστό σφάλματο. Δεν υπάρχει τεράστια βελτίωση. Στο περιφερειακό ταμείο όμω όχι. Γιατί? Ίσως γιατί ο Επίτροπος για τις κοινωνικές υποθέσεις είπε ότι αν ένας έλεγχος μηχανισμού δεν είναι ορθός, τότε σταματάμε τις προκαταβολές. Να, γιατί να μην κάνουμε λοιπόν το ίδιο και με το Περιφερειακό Ταμείο. Γιατί ο αρμόδιος επίτροπος διστάζει να σταματήσει τις πληρωμές λόγω του 3,7% ποσοστού σφάλματος που αυξήθηκε από το 3,2%. Τώρα δεν θα αναφερθώ σε όλες τις ειδικέ εκθέσεις, αλλά υπάρχει και μία για τα Ηνωμένα Έθνη. Στην περίπτωση έκτακτων δράσεων, υπάρχει λόγος να μπλέκεται να μπλέκονται Ηνωμένα Έθνη. Αλλά στις άλλες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη δίνουν χρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύοντας ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της δίνει τα χρήματα στην Ηνωμένα Έθνη, ε, αυτό είναι bypass. Δεν είναι αναγκαίο. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν τέτοια χρήματα να τα δίνουν κατευθείαν στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Συνεπώς εμείς ως φιλελεύθεροι εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί για την συμμετοχή μας όταν πηγαίνουν χρήματα στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε. Είναι η δουλειά των ίδιων των Ηνωμένων Εθνών, οπότε εμεί δεν βλέπω τη δουλειά έχουμε εκεί. Αυτές πρόεδρε ήταν κάποιες προκαταρτικές μου παρατηρήσεις όσον αφορά την φετινή απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> αγαπητέ κύριε Μούλδο, εξωγόμενο της ομάδας του της Άλτε. Κύριος Μπράντμπερν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ίσως να υπενθυμίσω την ε, τις παρομοιώσεις με το, την ταινία Casablanca όπου στο παρελθόν λέγαμε round up the usual suspects, να συλλάβουμε τους συνήθεις υπόπτους. Τώρα περισσότερο θα ανέφερα τη φράση play it again Sam, Ξαναπέξτε το Sam. Έχουμε αυτή την επαναλαμβανόμενη επανάληψη. Την αιτήσει αυτή η ερωτελεστία ε, δικαιολογιών γιατί υπάρχουν προβλήματα με την τελική απαλλαγή του προπολογισμού. Θέλω να αναφερθώ σε μερικά γενικά σημεία, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, συζητήσαμε ήδη και με, τον, με την κυρία Υπουργό και μετά από αυτά που ακούστηκαν, αναφέρθηκε το θέμα των ποσοστών σφαλμάτων για ορισμένε περιοχέ δαπανών. Ξέρουμε ότι περίπου 90% από τα σφάλματα προέρχονται από το επίπεδο των κρατών μελών. Η έκθεση όμως του κυρίου Φιέλνερ είναι απόλυτα έγκυρη, γιατί ο Κύριο Φιέλνερ τονίζει ότι η Κομισιόν δεν έχει κάνει αρκετέ προσπάθειες για να γίνει σαφές τα κρατημέλη, τα οποία δεν λειτουργούν καλά στην, στον έλεγχο αυτών των ταμείων, ότι πρέπει να πράξουν κάτι. Σύμφωνα με αυτό που λέει, ότι τα κρατημέλη έχουν προβλήματα τελικά <clears throat> με τις περιφέρειές τους, γιατί πολλές φορές οι τελικοί δαπάνοι γίνονται γίνεται στις περιφέρειες. Δεν μπορεί όμω η Κομισιόν να αποσύσει την ευθύνη τη και να τη μεταφέρει στα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν σφάλματα σε επίπεδο κρατών μελών. Άκουσα αυτά που είπε ο Επίτροπος σε σχέση με αυτά που θέλει να κάνει για να βελτιώσει την κατάσταση. Αλλά ανησυχώ ιδιαίτερα όταν έχουμε παραγωγή το θέμα των δαπανών στο Ταμείο Συνοχή για την αύξηση στο ποσοστό σφαλμάτων εκεί. Αν θέλουμε να πετύχουμε λύσεις χρειαζόμαστε και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό κυρώσεων που προφανώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεδομένης της σαφού αποτυχία και αστοχία μα στα θέματα αυτά και τη αύξηση στα ποσοστά ασφαλμάτων, δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτή την κατάσταση. Συμφωνώ με τον εισηγητή απόλυτα όταν λέει ότι η Κομισιόν πρέπει να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο στο να αναπτυχθούν κοινέ διατάξει για τα διάφορα ταμεία. Και πρέπει να είναι όσο το πιο αυστηροί αυτοί οι κανόνες όπως είπα προηγουμένως κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής. Και ανησυχώ επίσης και για τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου για το χαμηλό επίπεδο εκθέσεων της Κομισιόν. Το κοινόβουλιο δεν μπορεί να βασίζεται στις εκθέσεις της Κομισιόν για την απόδοση στα κονδύλια αυτά. Ζητώ λοιπόν να υπάρξει μια συστηματική ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων. Γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε πολλά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και από το Ελεκτικό Συνέδριο και τον κύριο Φιέλνερ. Και γιατί. Και το λέω αυτό εν, εν είδη κατακλείδος. Γιατί δεν συνεχίσαμε τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει στην πρώτη Επίτροπη Μπαρόζου του να υπάρχει ένας επίτροπος αρμόδιος για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και αν η Κομισιό θέλει να είναι σοβαρή για το να αντιμετωπίσει τα θέματα τα οποία ετέθησαν από τις διάφορες αυτές εκθέσεις πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο να εξασφαλίσει την σωστή αξιολόγηση των προγραμμάτων, τη σωστή χρήση των κοδηλίων και την πλήρη λογοδοσία για τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπράντμπορν. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να έχει ζητήσει το λόγο. Έχει κλείσει επόμενο ο γύρος στον ομιλητών. Κύριε Σιωμέτα θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν θέλετε να κάνετε και εσείς μια απάντηση, μια παρέμβαση που μορφή απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έλεγχαν σε αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικά σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ετέθη το θέμα του φρένου ασφαλείας για τα συστήματα αυτά. Δεν έχουμε καμία τέτοια δυνατότητα στο τωρινό πλαίσιο, αλλά μπορούμε να προτείνουμε αλλαγές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν με την ε, πρόορη ε, απελευθέρωση των ποσών από τα κράτη-μέλη και τη μελλοντική τους χρησιμοποίηση για, μέσα σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Αυτό δεν έτυχε υποστήριξη από τους συν-νομοθέτες. Μπορούμε να το επανεξετάσουμε αυτό όμως στα πλαίσια της προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο πολυετούς σχεδιασμού Μπορεί να συμπεριληφθεί και το θέμα αυτό λοιπόν στη συνολική εξέταση. Για την προχρηματοδότηση και μια ενδεχόμενη μελέτη για τα θέματα αυτά όπως είπα στην εισαγωγή μου πράγματι είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια ανάλυση των ενεργειών προχρηματοδότηση από το 2005 στο 2010. Το θέμα που τίθεται εδώ είναι ότι συνήθως η προ χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε επίπεδο σφαλμάτων όπως σε άλλες ενέργειες. Τα σφάλματα στην προχρηματοδότηση είναι συνήθως χαμηλότερα από τα σφάλματα για την ενδιάμεση χρηματοδότηση και τις τελικές χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το ελεκτικό συνέδριο <clears throat> ζήτησε να υπάρξει αλλαγή στη μεθοδολογία του και να εξαιρέσει την προχρηματοδότηση από τον έλεγχό του και να δώσει έμφαση μόνο στις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές μέσα στη διαδικασία δειγματοληψίας. αλλά συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι η προχρηματοδότηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως αυτή την οποία διαρχόμαστε είναι απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσει να δοθεί χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη μας σε σχέδια εν εξελίξη Αυτά λοιπόν τα οποία συμφωνήθηκαν κάτι διακέ, διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πώς θα αντιμετωπιστεί η προχρηματοδότηση στο δημοσιονομικό κανονισμό, όλα αυτά είναι μια συμβιβαστική λύση που θα μας βοηθήσουν και στις μελλοντικέ ενέργειες στον τομέα αυτό. Για την αντικατάσταση των σχέδιων η πρόταση για, το επόμενο, για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού σχεδιασμού είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιείται αυτή η αναδρομική προσέγγιση για την αντικατάσταση σχεδίων. Αν εγκριθεί λοιπόν αυτή η αλλαγή από τους νομοθέτες, από τα δύο σκέλη της νομοθετικής εξουσίας, αυτός θα είναι και ο κανόνας και προσβλέπω στην συνεργασία του Κοινοβουλίου για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Και θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Οι αιτήσει δηλώσεις τώρα. Η προσέγγιση την οποία προτείνει η Κομισιόν στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στο να έχουμε αιτήσεις διαχειριστικές δηλώσεις σε επίπεδο κρατών μελών και αφού και σε, ευρω... Ευρω... σε δηλώσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο που μπορούν εν καιρό να γίνουν εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα κράτη-μέλη μας διστάζουν πολύ να αντιμετωπίσουν να εφαρμόσουν αυτή τη μεθοδολογία. Προσβλέπω λοιπόν σε μια στενότερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο ώστε να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι, οι διατάξεις να μείνουν μέσα από τις τροπολογίες του δημοσιονομικού κανονισμού για τις αιτήσει <clears throat> συνόψεις η τωρινή νομοθεσία δίδει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πούν εάν συμφωνούν <clears throat> ή όχι να δημοσιοποιήσουν αυτές τις συνόψεις ή όχι και κάποια κατημέλη συμφωνούν με αυτό. Όλες, όλα τα κατημέλη συμφωνούν με αυτό και μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο μπορεί αυτό να είναι μια πραγματικότητα. Τέλος, για τις ε, χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις του EFF, EFSF ή του ESM. Η νομοθεσία για το ESM είναι σαφής, λέει ότι, ότι το ελεκτικό συνέδριο ή ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου θα συμμετάσχει ως μέλος στο πάνελ ελέγχου και τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν από το ESM θα είναι αντικείμενο λογιστικού ελέγχου με πλήρη συμμετοχή του ελεκτικού συνεδρίου. <coughs> Αυτό το σημαντικό λοιπόν στοιχείο θα επιτρέψει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια για τη χρήση αυτών των διευκολύσεων και σε σχέση με το θέμα των των ε, διαρθωτικών πόρων έναντι το, του κοινωνικού ταμείου, εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το 2010 ήταν το πρώτο έτος όταν όλα τα προγράμματα στον τομέα της συνοχής ξεκίνησαν. Τα ποσά λοιπόν αυτά τα οποία <clears throat> έχουν δαπανηθεί για την πολιτική συνοχή σχεδόν διπλασιάστηκαν έναντι των προηγουμένων ετών ενώ το ποσοστό των σφαλμάτων αυξήθηκε από 5,8 σε 7,6 αλλά το επίπεδο σφαλμάτων ήταν ε, πολύ χαμηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά ήταν στην εκκίνηση και δεν είχαν φτάσει την πλήρη του ταχύτητα, μπορούμε να περιμένουμε ότι τα επερχόμενα έτη θα μπορέσουμε να μειώσουμε το επίπεδο των σφαλμάτων και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Εμείς χρησιμοποιούμε ενεργά τις κυρώσεις αυτές και όπως ανέφερε και ο εισηγητής, δεν διακόψαμε, δεν, αναστήλαμε πληρωμές για περιφερειακά ταμεία το 2010, αλλά στην αρχή του ενεστώτος έτους η Κομισιόν αποφάσισε να αναστείλει ένα μεγάλο αριθμό κονδυλίων δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά επιδοτήσεις προς τις περιφέρειες της Ευρώπης Εφαρμόσαμε λοιπόν αυτό το μηχανισμό κυρώσεως με πολύ σοβαρό τρόπο και όταν εντοπίζονται σφάλματα επιμένουμε να εξασφαλιστεί η διόρθωση αυτών των σφαλμάτων και επιβάλλονται κυρώσεις υπομορφή αναστολής ή διακοπής των πληρωμών σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται όμως χρόνος μέχρι να κατανοήσουν και οι τελικοί αποδέκτες των κονδυλίων αυτών ότι μας ενδιαφέρει πολύ και είμαστε σοβαροί στην εφαρμογή του μηχανισμού αυτού κυρώσεων και μόνο τότε θα υπάρξουν βελτιώσεις. Για τις ανακτήσεις. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν προχωρούν αυτή τη στιγμή σε έναν έλεγχο σε μια σειρά κρατών μελών σε σχέση με τις ανακτήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα απεικονίζονται και στην ετήσια έκθεση του Γενικού Διευθυντή για το 2011. Και μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους θα παρουσιάσουμε τα συνολικά πορίσματα αυτών των λογιστικών ελέγχων και θα συμπεριλαμβάνουμε και τις προτάσεις μας για το τι μπορεί να βελτιωθεί στο σύστημα ανάκτησης στα κράτη-μέλη μέσα στο τωρινό νομικό πλαίσιο βέβαια γιατί οι προτάσεις που έχουμε κάνει θα εφαρμοστούν πλήρως από το 2014 μονάχα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μοναχά το τωρινό πλαίσιο όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ώστε Ελπίζω ότι έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σε σχέση με την, ε, ε, επίσης με την ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Υπάρχει και το θέμα του δημοσιονομικού κανονισμού. Προτείνουμε να δημιουργήσουμε καταπιστεύματα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πρόοδος λοιπόν στα θέματα αυτά και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών για τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω ότι τώρα έχω καλύψει όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν και αφορούσαν την Κομισιόν και όπως είπα και στην ε, <clears throat> αρχική μου παρέμβαση είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια επιστολή, μια γραπτή επιστολή που περιλαμβάνει, θα περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες δράσεις που θέλει να αναλάβει η Κομισιόν στο εγγύς μέλλον για να αντιμετωπίσει τους τομείς προτεραιότητας που έχουν υπογραμμιστεί από τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα, για να κλείσει το θέμα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Φέλνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Σεμέτα. Πρέπει λοιπόν να πω ότι απαντήσατε σε πάρα πολλά σημεία και ο τρόπος με τον οποίο απαντήσατε ε, αποδεικνύει και την, το πολύ καλό κλίμα που επικράτησε μέχρι τώρα στη συνεργασία μας. Αλλά ένα πράγμα θέλω να πω ότι προσβλέπω και στη γραπτή σας απάντηση γιατί αυτό θα αποδείξει ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να προχωρήσει, να προσυπογράψει αυτά τα οποία είπε. Ε, πολλά από αυτά που είπατε στην ομιλία σας ε, πάρα, πολλές, ε, καλές απαντήσεις δώσατε. βεβαίως, ορισμένα θέματα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ας πούμε για το θέμα της πολιτικής ευθύνης των ε, ετήσιων προγραμμάτων ε, πεπραγμένων. Και επίσης ε, πρέπει να συζητήσουμε και με τους αδέλφους το ποια είναι μια λογική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω και βεβαίω πρέπει να συνεχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Γκάια για να δω πού μπορεί να προκύψει προστιθέμενη αξία ή που πιστεύει θέμενη αξια απλά επαναλαμβάνεται κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον το ότι η Κομισιόν αναζητά ένα μοντέλο όσον αφορά το θέμα της ευθύνης. Είμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη να ε, ενημερώσει τον Επίτροπο. Εγώ προσωπικά ε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο Επίτροπος δεν ήθελε να απογράψει ότι εγώ ενημερώθηκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε ε, το πώς μπορεί να επικρατήσει μια λογική ισορροπία. δεύτερη καλή είδηση και αυτή ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Πριν από 10 λεπτά το γραφείο μου πήρε ένα email από τον κύριο Όσενμπορκ. Δεν ξέρω ε, κατά πόσον ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της Δανίας ή Υπουργός που είπε ότι τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να συζητήσουν μαζί μας το θέμα του πώς ε, εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη το θέμα της ε, επιμερισμένης διαχείρισης. Ίσως να ήταν ο κ. Μπράτπορ ο οποίος ε, διαχείρισε, ε, αντέδρασε. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν ήθελε να συζητήσει με τους ευρωβουλευτές το θέμα του ποσοστού σφάλματος. Αλλά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης ένα από τα κράτη-μέλη ε, στο οποίο επευθυνθήκαμε είπε ότι είναι πρόθυμο να συζητήσει το θέμα και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια καλή αρχή. Και τώρα περιμένουμε τους άλλους δύο, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς, να δούμε αν θα συνεχίσουν να έχουμε ευχάριστες ειδήσει. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Γκάια είπε ότι μπορεί να υπάρξει ε, κάποιο διάλειμμα στο θέμα των ε, χρηματοπιστωτικών μέσων. Βεβαίως ε, μπορεί να μας προσφερθεί μια ευκαιρία να επανέλθουμε στα, στα μέσα της χρηματοοικονομικής τεχνικής. Αυτό δεν είναι άλλο θέμα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προχρηματοδοτήσεις, ο κύριος Γκάια έχει απόλυτα δίκιο ότι τώρα έχουμε και πολιτική ευθύνη για αυτό το θέμα. Ζητάμε πράγματα, ε, η Κομισιόν ανταποκρίνεται και μετά γεμάζεται πολύ δύσκολο να ασκήσουμε κριτική. Βεβαίως το να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από αυτά τα κονδύλια ως απάντηση στην κρίση, αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι ε, σημαντική η ταχεία εκτέλεση και οι προχρηματοδοτήσεις είναι εξίσου σημαντικές. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει βέβαια να διεκδικούμε την εκτέλεση χάνει και μόνο της εκτέλεσης ε, ούτε να χρησιμοποιούμε τις ε, προχρηματοδοτήσεις για απλά να χρησιμοποιούμε ε, αυτό το μέσο στις εξωτερικές σχέσεις. Γιατί αν δούμε τα στοιχεία θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένους τομείς ε, υπήρξε βελτίωση απλά και μόνο επειδή υπήρξαν προχρηματοδοτήσεις. Και στις ε, προχρηματοδοτήσεις δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος σφάλματος όπως στις τελικές πληρωμές, σε καθαρίσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τέταρτο. τα αναδρομικά προγράμματα. Και ο λόγος που δεν το ανέφερα είναι ακριβώ ο ίδιος που ανέφερε και η Κομισιόν. Δηλαδή αυτό γίνεται δική μας πολιτική ευθύνη να μεριμνήσουμε, να πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε αναδρομικά προγράμματα στο τελικό ε, νομοθετικό πλαίσιο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει ε, ευρωπαϊκή προστέμενη αξία ε, σε αναδρομικά προγράμματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά και χαίρομαι που το αναφέρει αυτό και η Κομισιόν. Ο κύριος Μούλντε είπε κάτι σχετικά με τη δημοσίευση των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ συμφωνώ, λογικό μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει, αλλά γιατί όχι. Αν υπάρχει κάποια αξία, αν αυτό εξυπηρετεί, γιατί όχι, να δημοσιεύονται οι εκθέσεις. Και τέλος, το θέμα των κυρώσεων, του μηχανισμού κυρώσεων. Άκουσα τον Επίτροπο που μίλησε για το μηχανισμό κυρώσεων και είπε ότι ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για τα κρατη για να κατανοήσουν την ε, αποτελεσματικότητα στην διακοπή των ε, ε, πληρωμών. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και γι' αυτό το συζητήσαμε. Γίνεται συνεχώς λόγο για αναχαιτήσεις, για διακοπές. Πάντως εγώ προσβλέπω στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανακτήσεις. Γιατί είναι ενδιαφέρον όταν γράφει κανείς, όταν συντάσσει μια έκθεση, τότε διαπιστώνει ότι πρέπει να έχει και άλλες πληροφορίες ε, ότι αυτές θα βοηθήσουν και είναι λυπηρό ε, το ότι το μέλλον είναι πιο ενδιαφέρον από το παρελθόν ε, και από ό,τι φαίνεται ε, οι πιο ενδιαφέρουσε εκθέσει επίκυνται ακόμα. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που μας είπατε θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Αυτά είχα να σας πω και σας παρακαλώ να μου καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή είναι σαφές νομίζω το χρονικό διάστημα, η κατάσταση απολογιών μέχρι τις 5 Μαρτίου, η ψηφοφορία 26 Μαρτίου. Κλείνει και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο που ήταν πρόθυμος ε, να απαντήσει ε, στις ερωτήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ για την επόμενη συνάντησή μας στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Äh, Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο υπερθμών που πρόκειται για την απαλλαγή του 8ου, 9ου και 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, εισηγητής ο κ. Μάρτιν Ερενχάουζερ. Και εδώ οι τροπολογίες μέχρι την 5η Μαρτίου ε, και η ψηφορία στις 26. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να περιμένουμε λιγάκι μέχρι να φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν. Κοιτάξτε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Στις 6.30 πρέπει να τελειώσουμε. Οι συζητήσεις παρακαλώ να γίνουν εκτός της αίθουσας. Ich Θα προσπαθήσω ε, όσο το δυνατόν να κάνω αυτό που μου ζητάτε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το θέμα της απαλλαγής. Εγώ θα πρότεινα να δοθεί η απαλλαγή για το 2010. Δεν υπήρξε κάποιο έκτατο γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε αντίθετη πρόταση. Αυτό όμως το ισχύει πάντα είναι αυτά τα σταθερά στοιχεία τα οποία ανέφερε ο κύριος ε, Μούλτερ για την Κομισιόν. Για το θέμα των Evergreens λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο να κρατηθεί μια ε, σόφρον στάση σε σχέση με την αντιμετώπιση των άλλων θεσμικών οργάνων και έτσι αυτά τα λεγόμενα evergreens θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Μέχρι τότε είναι χρήσιμο να προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση του Ταμείου Ανάπτυξης στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι υπάρχει μια σημαντική δυνατότητα να επιτευχθεί αυτό μέσα στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014 ε, μέχρι το 2020. Βέβαια υπάρχει και ένας περαιτέρω λόγος που είναι η εκπνοή της Συμφωνίας του Κοτονού. Θα πρέπει να εξασφαλίσει λοιπόν η Επιτροπή μας τη δυνατότητα να ασκηθεί η καταληπίεση προς το Συμβούλιο ώστε το έτοιμο αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να γίνει δεκτό. Ένα άλλο θέμα είναι πάντα το ποσοστό σφαλμάτων για το 2010 ήταν 3,4%. Ξεπερνάει βέβαια το κατόφλι του 2%. Η Κομισιόν έχει εκφράσει την εντύπωση ότι αν δει κανείς ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δει ολιστικότερα τα θέματα, έχει μείνει σταθερό το επίπεδο των σφαλμάτων, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ο στόχο τη Επιτροπή μα και πρέπει να το πω εκπεφρασμένο. Στόχο δεν είναι σταθερό το ποσοστό σφαλμάτων, είναι να μειώνεται το, σφάλμα, το ποσοστό σφαλμάτων και οι ενέργειε τη Κομισιόν δεν το έχουν επιτύχει αυτό. Επίση για τα το υπολοιπόμενο επίπεδο σφαλμάτων, λέει η Κομισιόν ότι παραμένει κάτω από το επίπεδο σημαντικότητα του 2%, αλλά η Κομισιόν δεν μπόρεσε να μα δώσει σαφεί δείκτε ή να πει με σαφή τρόπο πώς καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει να μας δώσει και τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε ποια είναι και η οικονομική σημασία όλων αυτών των υπολοιπωμένων σφαλμάτων και ελπίζουμε ότι μέχρι το 2013 οι δείκτες για τα υπολοιπόμενα επίπεδα σφαλμάτων θα έχουν ε, εφαρμοστεί πλήρως. Εν τάχει για το σύστημα παρακολούθησης και υποπτίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά από συστήματα για την εποπτεία αυτή αλλά για μας είναι σημαντικό να έχουν μια ορατότητα και μια διαφάνεια αυτά τα συστήματα ε, παρακολούθησης. Έχουμε πάρει αυτό το οποίο για πολύ καιρό ζητούσαμε την Κομισιόν μια έκθεση για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάπτυξη. Αυτό βέβαια δεν είναι επιτυχία, έπρεπε να είχε γίνει ήδη στο παρελθόν. Ένα άλλο Everton, μια άλλη μόνιμη απέτηση είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού και νομίζω ότι αυτό το οποίο απαιτούμε είναι να υπάρξει πλήρης έλεγχος από την σχεδίαση μέχρι την εφαρμογή, μέχρι την τελική αξιολόγηση. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μείωση των ποσοστών σφαλμάτων και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συνολική μεταρρύθμιση. Είδαμε σε πολλές χώρες όπως και η ΑΕΤ πόσο σημαντικό είναι το εργαλείο αυτό για να μπορέσει κανείς να οικοδομήσει μια μεταρρύθμιση και να εξασφαλίσει την πρόοδο στα μέρη αυτά και είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι έχει γίνει με ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και αυτό απαιτεί και ένα σταθερό διάλογο με τις χώρες με τις οποίες εμείς έχουμε ε, αναπτυξιακές ενέργειες. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε είναι το λεγόμενο, η λεγόμενη διευκόλυνση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εγώ προσπάθησα να το δω αυτό το θέμα λίγο πιο ε, προσεκτικά κατά την εντύπωσή μου, παραμένουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ελέγξει καλύτερα το ελεκτικό συνέδριο. Ταμιακέ ροέ, καταρχήν, από, την από τα κράτη-μέλη προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα. Κατά την άποψή μου αυτό είναι μια πολύ μακροχρόνια διαδικασία και είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία όπως παραδοσιακά το τραπεζικό απόρριτο και γι' αυτό η πρότασή μας είναι να συντάξει μια ειδική έκθεση του Ελεκτικό Συνέδριο για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της μεταβίβασης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων σε διάφορες ε, τράπεζες. Τέλος, να πω κάτι σε σχέση με την αποστολή μας στην ε, ε, IT για την ανακουφιστική βοήθεια που θέλουμε να δώσουμε στην IT. Έχουμε σε στόχο να έχουμε μια μεταβατική βοήθεια η οποία γεφυρώνει μεταξύ ανακουφιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας το κενό το οποίο δημιουργείται και έχουν ε, προταθεί τα μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο συντονισμό για τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας πω. Θα τα ευχαριστήσω και την Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συνεργασία που έχουν, ε, μου έχουν προσφέρει. Ήταν πολύ ε, ήταν χωρίς καθόλου προβλήματα αυτή η συνεργασία. Θα ευχαριστήσω λοιπόν όλα αυτά τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γκάια έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Αποκινούμε τον εισηγητή. Είμαστε λιγάκι περισσότερο πλέον απογοητευμένοι για το ότι η Κομισιόν ε, δεν κατόρθωσε να εγγράψει πλήρως ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, στον προϋπολογισμό. Αυτό αποκλείεται να γίνει στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 και είναι ένα θέμα, είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα της δικής μου της πολιτικής ομάδας που δεν γίνεται αποδεκτό. Και το πληρώνουμε με το ότι ε, υπάρχει έλλειμμα σαφήνειας ε, και διαφάνειας. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λυπούμεθα πάρα πολύ γι' αυτό και κατόπιν τούτου συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή. Συμφωνούμε επίσης με τον εισηγητή για το ότι τα λάθη, τα σφάλματα που υπάρχουν στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων ε, προκαλούν ανησυχία και στηρίζουμε πλήρως ε, τα μέτρα τα οποία προτείνονται στον τομέα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα ποσοστά σφάλματος. Επίσης ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει κάποια διαφορά στα ποσοστά σφάλματος. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει σε μια διαφορετική προσέγγιση διαφορετική ετήσια προσέγγιση, ε, ενώ η Κομισιόν εξετάζει το θέμα αυτό ε, σε, μια, ε, σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα χαιρόμασταν αν τελικά προέκυπτε ένας μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε τη δυνατότητα σύγκρισης των παρατηρήσεων στο μέλλον. Επίσης, συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή για το ότι στον τομέα της δημοσιονομικής βοήθειας κάτι πρέπει να γίνει. Ο κύριος ε, παρέπεμψε στην αντιπροσωπεία για την IT. Ε, αυτό είναι αλήθεια. 62 εκατομμύρια στον, ε, να δώσουμε στην Αιτή και να γραφούν αυτά στον προϋπολογισμό της έτσι ώστε μετά το σεισμό να ανοικοδομηθεί η διοίκηση. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφραστεί επανειλημμένα το αίτημα να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός, να ενισχυθεί η βοήθεια. Αυτό όμως, αν γίνει, τελικά πρέπει να συνδυαστεί με καλύτερη διαφάνεια ε, και ε, πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τελικά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω το εργαλείο αυτό. Εκείνο το οποίο επίσης ε, χαιρετίζουμε είναι το εξής, ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιου είδους ε, πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενοι. Αν θέλετε αυτά είχα να πω στην ε, έκθεση, για την έκθεση αυτή Κατά τα άλλα, ε, θα ήθελα να ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, επόμενος, ο συνάδελφος κ. Χολμάια. Ή συνάδελφος, η συνάδελφος, με κυρία Χολμάια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο εισηγητή για την πλήρη και ενδελεχή και εξισορροπημένη έκθεση την οποία μας παρουσίασε. αντιμετωπίζει φυσικά την ε, βασική προβληματική την οποία έχουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην Επιτροπή μας για τα θέματα της ε, ε, αρρωγής στον προϋπολογισμό. Έχω ήδη θέσει μια σειρά ερωτήσεων στον αρμόδιο επίτροπο Μπίμπαλκ για θέματα τα οποία εμείς υποστηρίζουμε και προτείνουμε εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαίτερα για το θέμα της διαχείρισης των διεργασιών που θα πρέπει να συμπεριληφθεί πιο στενά μέσα στην, ε, στον έλεγχο της χρηματοδότησης και φυσικά και να συνοδεύεται με το θέμα της, ε, του ελέγχου της τακτικότητας αυτής της χρηματοδότησης και να εξετάσουμε φυσικά κατά πόσο οι τοπικές αρχές στις οποίες δίδεται αυτή η αρρωγή είναι σε θέση πράγματι να εκτελέσουν τα σχέδια για τα οποία χρηματοδοτούνται και δεν πηγαίνουν σε άλλα κανάλια και αυτά, τα, κονδύλια αυτά. Επομένως είναι απαραίτητο για το θέμα του, της αρρωγής στο προϋπολογισμό ε, να παραμείνουμε επάγρυπνοι γιατί αλλιώς ένας από τους σημαντικούς μηχανισμούς της αναπτυξιακής βοήθειας ξεφεύγει από τους ελέγχους μας και αναρωτιέμαι γιατί δεν δίνουμε αρκετή έμφαση εδώ πέρα στο θέμα της διαχείρισης. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερους μηχανισμούς, ε, ενδεχομένως να εξετάσουμε και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων μηχανισμών ελέγχων με τις χώρες αυτές, ώστε να επιτύχουμε το στόχο που επιθυμούμε. Συμφωνώ την άποψη ότι θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό και αυτό νομίζω το να γνωρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες να ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και στον προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια θα γίνει ούτως ή άλλως με την ε, εκπνοή της συνθήκης της Κοτονού το 2020, αλλά είναι μια πάρα πολύ μακρά ιστορία για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάντα, ότι έχουμε διαφορετικά καλάθια τα οποία πρέπει να ελέγχουμε με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Είναι χρήσιμο να τα συνενώσουμε όλα αυτά για να υπάρξει μια πλήρης ευθύνη και να μην μπορεί κανείς να υπερκφεύγει λέγοντας εγώ ελέγχω το πρώτο καλάθι και όχι το δεύτερο ή το τρίτο καλάθι. Αυτό δεν κάνει πιο αποδοτική αυτή τη διαδικασία και ίσως και τα κάτι μέλη θα πρέπει να σκεφτούν καλύτερα πόσο αποδοτικό είναι το κάθε κράτος να μπορεί να συνεχίζει αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα προγράμματα άλλων κρατών και παράλληλα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυξάνει την αποδοτικότητα των προγραμμάτων αυτών και πρέπει να αποτελέσει και πάλι αντικείμενο <clears throat> συζητήσεων. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τα σχεδιά, σχεδιά της στα σημεία 64 και 65. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Εδώ αναφέρεται η περίπτωση ενός ε, μη κυβερνητικού φορέα Αναφέρεται το θέμα λοιπόν της ανάγκης να υπάρξει μια ανάκριση ή ακόμα και αγωγή στην περίπτωση αυτή διότι υπάρχει υποψία διαφθοράς και έκπλησης χρημάτων. Εδώ θα ήθελα να έχω και καλύτερες πληροφορίες, πιο νοπές πληροφορίες για το κατά πόσο είναι έγκυρη και αξιόπιστη, είναι έγκυρος και αξιόπιστος αυτός ο, οργανισμός ή η μη ή οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φυσικά δεν θέλουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ένα άλλο σημείο κριτικό αφορά το σημείο 68 μέχρι το σημείο 72 Πρόκειται για ορισμένα σημεία τα οποία βρίσκονται πραγματικά εκτός της δυνατότητας ελέγχου μας. Τα επιμίσθια, τα μπόνους παραγωγικά του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται η <clears throat> αποπληρωμή των χρεών για, το, για τα υψηλά επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια σε σχέση με άλλους πιστωτές. Εγώ έχω πραγματικά θέσει το ερώτημα του κατά πόσο όλα αυτά εμπίπτουν στην διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου μέσα στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι αυτά τα σημεία 68 38 μέχρι 72 σε κάποιο σημαντικό βαθμό εκφεύγουν από τις αρμοδιότητές μας και θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα αν έχει νόημα να συζητούμε με τέτοια στοιχεία. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απαλλαγή της Κομισιόν και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόλμα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα επιμίστια της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρίσκεται στο ακραίο, στο ακρότατο όριο αυτού που λέμε αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο? Ο Όλες Σμιτ έχει το λόγο. Thank you, Mr. Uh, I was in... Ευχαριστώ. Ήμουνα στην Ζάμπια, κύριε. Την προηγούμενη εβδομάδα και σχολίασαν εκεί μία έρευνα σε σχέση με τη διαφθορά. Οι πολίτες στη Ζάμπια, λοιπόν, λένε ότι οι δικοί τους, οι βουλευτές, οι πολιτικοί είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι μηνύματα στέλνουμε από την Επιτροπή μας σε σχέση με τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς στις διάφορες ε, χώρες όπου στέλνουμε και βοήθεια. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και συμφωνώ περίπου με τα πάντα. Όμως, ό,τι λέμε για το δικό μας ε, τον προϋπολογισμό δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Τώρα υπάρχει κάτι που μου αρέσει να ακούω. Τα επιχειρήματα δηλαδή τη δημοσιονομική στήριξης. Κοιτάξτε, είναι επικριτική η έκθεση στην δημοσιονομική αυτή στήριξη και μπορώ να το καταλάβω. Από την άλλη όμως, αν θέλουμε οι κυβερνήσεις στις διάφορες χώρες όπου θέλουμε την βοήθειά μας να είναι πιο υπεύθυνε και εφόσον έχουμε έλεγχο και εποπτεία Νομίζω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Καταλαβαίνω τα προβλήματα, όμως θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα για τα επιχειρήματα, γιατί αν μιλήσετε με τους ανθρώπους αυτές της ε, υπονάπτυξη χώρες, ιδιαίτερα τις πολύ φτωχές χώρες, για αυτούς είναι φυσικά μια τεράστια πηγή, πολύ σημαντική, αλλά χρειάζεται έλεγχο. Βεβαίω και έχουμε ευθύνε γι' αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ο έλεγχος που γίνεται και από τις ευρωπαϊκές αρχές στις Βρυξέλλες αλλά και επί τόπου, ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τα επιχειρήματα. Τα άλλα πράγματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ αυστηροί με αυτά και να προστατεύουμε όσους μας δίνουν πληροφορίες, τους whistleblowers, είναι ακριβώς οι πληροφορίες και η στήριξη αυτών που τολμούν να αποκαλύψουν πράγματα. συμφωνώ με τη διαδικασία Παρισάκρα και την, έτσι ώστε να υπάρχει εξοπιστία. Ήμουν στο Μπουζάνο που συζητήθηκε και εκεί η επάρκεια της βοήθειας τον Δεκέμβριο. Είχαμε την εισαγωγή της εταιρική σχέσης όχι μόνο με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο που και αυτό είναι ζωτική σημασία. Τελικά κύριε Γκάιερ. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δικιά μας αναπτυξιακή βοήθεια είναι μεγάλη. Είμαστε αυτοί που δίνουμε την μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ευτυχώς δεν είναι η κύρια πηγή ε, εσόδων για τις περισσότερες ε, χώρες. Οι επενδύσεις είναι όλο και πιο σημαντικές. Κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό η δικιά μας η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αναθεωρηθεί βάσει αυτής της νέας πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Πάντως, τον συγκεκριτή πιστεύω ότι είναι μια καλή έκθεση και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τη στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σμίτ. Επόμενη κυρία Αγιάλα Ζέντα. Ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτά που μόλις ακούσαμε, για τη δημοσιονομική στήριξη. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα να σας πω ότι όντας επικριτικοί, όπως είμαστε συνήθως, και με κάθε προσοχή που προχωράμε στη δημοσιονομική αυτή στήριξη, όμως να την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Μαυριτανία. Και εκεί ακριβώς κι εγώ Ζήτησα να ενημερωθώ για τα προβλήματα, γιατί υπήρξε ε, το πραξικόπημα και τις επόμενες μέρες απευθείας πάγωσε όλη αυτή η δημοσιονομική βοήθεια, εκτός από το ανθρωπιστικό σκέλος. Και αυτό οδήγησε σε καθυστέρηση ενός έτους προκειμένου να ξαναρχίσουν σημαντικά προγράμματα που χαθήκαν. Όλοι οι υπάλληλοι πάντως της αντιπροσωπείας μας εκεί το είπαν. Η δημοσιονομική αυτή στήριξη έπρεπε βέβαια να υποβληθεί σε περιορισμούς εφόσον υπήρξε πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας έπρεπε να σταματήσει η χρηματοδότηση. Η Μαυριτανία πάντως αντιμετωπίζει και πρόβλημα του δικαστικού της συστήματος το γεγονός λοιπόν το να μπορέσει να προχωρήσει η δημοσιονομική στήριξη είχε σαν αποτέλεσμα να μπορούν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν λόγο ή τέλος πάντων να μπορούν κάπως να μιλήσουν για αυτά που βλέπουν στη χώρα, να βοηθήσουν και να συστήσουν πράγματα στις τοπικές αρχές. Άλλου είδους ε, βοήθεια δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, δεν δίνει το δικαίωμα λόγου ε, των υπαλλήλων μας πάνω στο σύστημα, το δικαστικό ή άλλο των κυβερνήσεων. Οπότε, λαμβάνοντα υπόψη όλα όσα λέει ο εισηγητής για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, συγχρόνως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό το γεγονός, ότι πρόκειται για ένα μέσο πολύ χρήσιμο που έχουμε στη διάθεσή μας ω Ευρωπαϊκή Ένωση και που μας δίνει το δικαίωμα άποψης για τα διαρθρωτικά συστήματα των χωρών, προκειμένου να είμαστε δηλαδή πιο απαιτητικοί για να πετύχουμε βελτίωση της κατάστασης επιτόπου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Κυρία Αγιάλα Σέντερ. Κάποια ερωτήματα τα οποία μπορεί να θέλει να αντιμετωπίσει και η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε κύριε Ισηγητά, Θα μιλήσω γερμανικά εφόσον είναι τόσοι πολλοί Γερμανοί βουλευτέ παρόντε και ελπίζω θα έχω την επίοικια των άλλων. Είναι πολύ περισσότερο, λέει ο πρόεδρο, από όσου βλέπετε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή ο οποίος προτείνει την ε, απαλλαγή και ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολύ επικοδομητικά τα θέματα αυτά στην έκθεσή του. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εμείς συμφωνούμε απλήρως με πολλές από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλά μέτρα έχουμε ήδη ξεκινήσει να θέτουμε σε εφαρμογή. <clears throat> Δεν ε, μπορούμε τώρα να σας τα παρουσιάσουμε πλήρως, ίσως σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσαμε να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία, ίσως για το θέμα της ε, δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσατε να έχετε μια ακρόαση στην οποία θα είχαμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε πώς ακριβώς ε, λειτουργεί αυτό το σύστημα και κάποια πράγματα ίσως θα μπορούσαν να σας εκπλήξουν. Σαν παράδειγμα για το 2011, συγγνώμη, για το 2011 υπάρχουν σημαντικά ποσά του ΕΤΑ τα οποία δεν μπόρεσαν να εκταμιευθούν γιατί οι προϋποθέσεις στις χώρες αποδέκτριες δεν, δεν ε, πληρούνται. Μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι κακό, ότι δεν υπήρξε η εκταμείευση αυτών των κονδυλίων. Από την άλλη μεριά όμω βλέπετε ότι εμείς είμαστε πολύ αυστηροί με τις προϋποθέσεις εκταμείευσης και όπως σας είπα το 2011 υπήρξαν σημαντικά ποσά τα οποία δεν αποδόθηκαν γιατί οι κυβερνήσεις με τις οποίες ε, θα συνεργαζόμασταν δεν εκπλήρωσαν τις προϋποθέσεις παρά το γεγονός ότι ζητήσαν να υπάρξουν αυτά τα ποσά. Έρχομαι τώρα σε αυτά που λέει ο εισηγητής. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο 2020 για, να δούμε τα λεγόμενα evergreens, τα μόνιμα αυτά θέματα να επιληθούν. Σε πολλά από αυτά έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε και έχουμε κάνει κάποιες πρόοδους, ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα επισητούσε το Κοινοβούλιο, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το 2020 για να τελειώσουν τα προβλήματα αυτά, τα evergreens, τα μόνιμα αυτά προβλήματα. Επίσης για το ποσοστό σφαλμάτων που αναφέρθηκε, εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ε, λεπτομεριακή και εμπεριστατωμένη μελέτη για να δούμε πώς προκύπτουν αυτές οι διακυμάνσεις στο ποσοστό των σφαλμάτων, πώς μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη επιμέτρηση αυτών των σφαλμάτων. Σε συνεργασία λοιπόν με το ελεκτικό συνέδριο έχουμε κάθε, στόχο, κάθε συμφέρον να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Πώ, παραδείγματο χάρη, όταν έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο να μειώσουν τα σφάλματα, μερικέ φορέ βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των σφαλμάτων. Και συμφωνούμε απόλυτα για το θέμα αυτό. Κάτι ακόμα για την ε, δημοσιονομική στήριξη και πάλι θα ήθελα να κάνω. <clears throat> Ήδη και το ελεκτικό συνέδριο έχει δεχθεί ότι είναι σημαντικό στοιχείο η δημοσιονομική στήριξη και ότι έχουμε επιτυχεί σημαντική προόδο σε διάφορους τομείς και στην εκτίμηση των κινδύνων και επίσης και για τα κριτήρια επιλεξιμότητος τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει να πάρει ένα κράτος δημοσιονομική στήριξη. Έχουμε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση όπου προτείνουμε να υπάρχουν και περαιτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας, παραδείγματος χάρη η διαφάνεια και ο έλεγχος του προπολογισμού στην χώρα η οποία είναι ο εταίρος μας, μόνο όταν έχουν εξασφαλιστεί από τον δημόσιο χώρο, από το κοινοβούλιο της χώρας αυτής, τότε η χώρα αυτή θα μπορέσει να πάρει αυτά τα, αυτή τη δημοσιονομική στήριξη στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε θα βελτιώσει και τη διαχείριση αυτών των δημοσίων κονδυλίων Επίσης, θεωρούμε ότι η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να λειτουργήσει μονάχα όταν ε, έχει βελτιωθεί και η διοικητική δομή. Γιατί με τον τρόπο αυτό όχι μονάχα βελτιώνεται η αποδοτικότητα της ε, δημοσιονομικής στήριξης, αλλά και η όλη ποιότητα της διαχείρισης στις χώρες αυτές. Και αυτό έχει φανεί από την εμπειρία μας και γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει μαζί με, τα, με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς να αναπτύξουμε εργαλεία μέτρησης της αποδοτικότητας ώστε να είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε και την αποδοτικότητα αυτών των μέτρων. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη δημοσιονομική στήριξη. Έχουμε ακολουθήσει μια σειρά από εσωτερικές κατευθυντήρες γραμμές και τις έχουμε κάνει σαφείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους. Μπορεί οποιοδήποτε να δει στο διαδίκτυο πόσο, ασ, πόσο αυστηροί είναι αυτοί οι κανόνες, δεν είναι μυστικές ρήτρε, όλοι τα γνωρίζουν, μπορούν ακόμα και στις χώρες που είναι αποδέκτες των κοδηλαίων να ελέγξει οποιοδήποτε τι ακριβώς γίνεται και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται αυτή η βοήθεια και έχουμε σε στόχο στο μέλλον να δημοσιεύουμε και τις συγκεκριμένε πληρωμές. Δεν γινόταν αυτό. Πήγαιναν τα ποντήλια αυτά στη χώρα που είναι αποδέκτη, παραδείγματο 50 ε, εκατομμύρια και κανεί δεν ήξερε τι γινόταν. Τώρα, από εδώ και πέρα, η κοινωνία των πολιτών, το κοινοβούλιο τη χώρα αυτή θα γνωρίζουν ότι έχουν αποδοθεί 50 εκατομμύρια στη χώρα αυτή και μπορούν, θα μπορούν να θέσουν πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, κλείνω για το θέμα αυτό. Δημοσιονομική στήριξη θα άξιζε πράγματι, όπω είπα, μια πλήρη ακρόαση Έρχομαι τώρα για το θέμα του ποσοστού σφαλμάτων. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από ενέργειες για, τα, για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων. Υπάρχει μια νέα πυραμίδα ελέγχου, υπάρχει ένα νέο σύστημα για την κατάρτιση στον τομέα αυτό και πιστεύω ότι σίγουρα θα βοηθήσουν στο να μπορέσουμε σταδιακά να έχουμε καλύτερο έλεγχο και λιγότερα σφάλματα. Υπάρχει πάντα μια βέβαια ένας, η ανάγκη ενός trade-off ενός συμβασμού μεταξύ καλύτερου ελέγχου και υψηλότερου κόστους ελέγχου. Και το έχουμε δει αυτό ήδη και με την περίπτωση των Ηνωμένων Εθνών ότι αν φτάσει πέρα από ένα ορισμένο όριο η αυστηρότητα των ελέγχων τελικά δεν επιτυγχάνει κανεί περισσότερα αποτελέσματα. Επομένω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αποδοτικότητα για, την, για τους ελέγχους αυτούς για το θέμα των Ηνωμένων Εθνών και τα κονδύλια που περνάνε από αυτά είναι ένα από τα evergreen, είναι από τα μόνιμα ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά λαμβάνουμε και εκεί τα απαραίτητα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν εν κατακλείδη να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί παρά τις διάφορες αμφιβολίες και ανησυχίες που εξέφρασε, υποστηρίζει την απαλλαγή. Πρόεδρος, ε, πριν κλείσουμε λοιπόν, θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Ε, Βλέπω η κυρία Κρέσλερ ε, ήδη ε, κοιτάει το ρολόι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας, γιατί ε, δεν θέλω αύριο να καθυστερήσουμε. Εντάξει, τότε θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα κάνω κι εγώ μια παρατήρηση αυτά που είπε η κυρία Χουλμάιρα. Σε τελική ανάλυση το όλο θέμα είναι πολιτικό. Πιστεύω βέβαια ότι το ερώτημα κατά πόσον το κοφόρο δάνειο μπορεί να θεωρηθεί πολιτικό εργαλείο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη χωρών, αυτό αμφισβητείται. Και εγώ πιστεύω λοιπόν ότι τέτοιου είδου γενική φύσεω παρατηρήσει θα έπρεπε να μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σε αυτή την έκθεση. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία λοιπόν. Όλα τα άλλα θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Κλείνει και αυτό το θέμα τη σημερινή διάταξη και πάμε στο επόμενο, στο 8. Πρόκειται για τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και καθεστώ που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συγγήτρια είναι η κυρία Κρίσλε. Θα ήθελα λοιπόν να τη δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πλατιάσω. Αυτή είναι η μόνη επιτροπή η οποία έχει ικανοποιητική βάση διαπραγματεύσεων. Εγώ έκανα λοιπόν το εξής. Αφενός ένα έγγραφο εργασίας ε, το οποίο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και αυτό αφορά την ε, ανάγκη μεταρρύθμισης ε, του κατσετικού. Αυτό σας το συστήνω να το διαβάσετε όλοι. Εκεί λοιπόν βλέπετε καταρχήν τους άμεσα θυγόμενους από τη μεταρρύθμιση και αναφέρονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι στους 10 οργανισμούς αλλά και τι κερδίζουν, ποιος είναι ο μισθός των απασχολούμενων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν πάρουμε ε, τους βουλευτές θα διαπιστώσετε ότι ένα τρίτο του προσωπικού κερδίζει περισσότερα από τους ευρωβουλευτές. Χαλάλι τους, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε σε αυτή τη δημόσια συζήτηση που κάνουμε. Έχουμε λοιπόν περίπου 25.000 που θα θυγούν από τη μεταρρύθμιση. Μετά σε ένα δεύτερο... Λοιπόν, αυτό το σημείο αναφέρεται και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το τι επιτυγχάνει αυτό το σχέδιο και τι όχι. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ αναφέρονται ε, κάποια μέτρα ε, αποταμίευσης, ε, κάποια προνόμια, τα οποία απαιτεί η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Και θεωρεί η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών ότι πρέπει να υπάρξουν τέσσερι μεταρρυθμίσει. Όμω η Ολομέλεια συμφώνησε μόνο σε ένα. Τα σημεία λοιπόν τα οποία απαιτεί η Επιτροπή δική μας ε, αλλά δεν τα ενέκρινε η Ολομέλεια. Ε, πρέπει να πω στην Επιτροπή ότι αυτό με χαροποίησε και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πάμε λίγο πιο πέρα από αυτά τα λίγα που απαιτεί η Ολομέλεια. Προσπάθησα επίσης ε, να σας ε, πω τι κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει. Διαπιστώνω λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος με το τι ακριβώς πρέπει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία. Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένας ε, απολογισμός, να προχωρήσουμε σε μια πραγματική μεταρρύθμιση. Τα θέματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας, δηλαδή αυτή που δίνει η σύγκρουση συμφερόντων. Για όλα αυτά δεν προβλέπεται τίποτα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, όμως εγώ εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω κάτι να προτείνω. Κατόπιν, στο πέμπτο σημείο προσπαθώ τις ε, τροπολογίες μου να τις αιτιολογήσω. Γιατί δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Ε, Παραδείγματο χάν οι μέρες επιστροφής στην πατρίδα. Θέλω να σε υπενθυμίσω ότι σε όλο τον κόσμο οι διπλωμάτες έχουν δύο μέρες. Εκτός από τους ε, εργαζόμενους στις Βρυξέλλες είχαν έξι, τώρα έχουν τρεις. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ε, πιο δύσκολο να έρθει κανείς από το τέλος του κόσμου και να ε, πάει στην πατρίδα του από το να πάει από τις Βρυξέλλες οπουδήποτε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Μετά, η ε, αντιστάθμιση με ελεύθερο χρόνο. Τι εννοώ. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το σχέδιο της μεταρρύθμισης δίνει τη δυνατότητα κυλιόμενου ωραρίου και αντιστάθμιση με ελεύθερο χρόνο. Αυτό είναι μια δυνατότητα που την έχουν όλοι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά του κυλιόμενου ωραρίου, αλλά τι γίνεται. Για ελεύθερο χρόνο μπορεί κανείς να προσθέσει 24 ημέρες. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι υπερορίες. Να το πούμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και να πούμε αυτό που υπάρχει και σε άλλες υπηρεσίες μία ημέρα το μήνα, κατά το μέγιστο. Φτάνει αυτό. Γιατί αλλιώς, αν δεν το ορίσουμε, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναπλήρωσης με ελεύθερο χρόνο που θα υπήρξε ποτέ. Ε, δεν μπορεί αυτό να παραμείνει ε, ως έχει. Πρέπει επίσης να καταθέσω και κάποιες άλλες ε, τροπολογίες. Προτείνω από το άντε 9 και πιο πάνω να περιλαμβάνονται οι υπερορίες στο μισθό. Και είπα ότι πλέον ε, δεν θα υπάρχουν ελεύθερες μέρες, αλλά ευέλικτο ωράριο. 18 ε, αργίες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές, 9 δεν είναι όμως εορτές που σημαίνει και αυτό προστίθεται ως αμοιβόμενες, ε, ε, αμοιβόμενε. άδεια. Εγώ προτείνω αυτές οι αργίες να περιοριστούν κατά τέσσερις για όλους. Τέσσερις λιγότερες. Τώρα, προτείνω επίσης ε, η αυτόματη προαγωγή, η ορίμανση όπως τη λέμε στα ελληνικά, να ε, είναι κατά 75 ευρώ το μήνα. Από δύο χρόνια μέχρι τρία χρόνια μέχρι την ΑΝΤΕ 12. 14.000 ευρώ το μήνα και από την άντε 12 η προαγωγή, η ορίμανση να έχει άμεση σχέση και με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στο ε ασχολούμαι με το παράρτημα 10 που αφορά συνεργάτες σε τρίτες χώρες, διπλωμάτες ή εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής κατάσταση. Οι συνεργάτες μας πολύ συχνά λείπουν από τη θέση εργασίας. Παίρνουν άδεια ή ελεύθερες ημέρες. Και έχω κάνει κάποια στατιστική για αυτές τις ελεύθερες ημέρες. Μέχρι και 59, 53 με 59 το χρόνο και έχω κάνει και κάποια σύγκριση με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και με το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει να σας πω, στη Γερμανία και στη Βρετανία, στα Υπουργεία Εξωτερικών τους, έχουν κατά ένα τρίτο λιγότερες ελεύθερες ημέρες, παρότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι μακριά από την πατρίδα τους. Βέβαια είναι δύσκολο να ε, περιορίσει κανείς αυτές τις ημέρες, αν δεν δει λιγάκι και της, ε, την ετήσια άδεια 30 μέρες στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία 30 μέρες άδεια. Άρα δηλαδή μιλάμε για 12 ημέρες ε, που προστίθενται, μέχρι τώρα δεν τις έχω αγγίξει, αλλά αν δεν τις αγγίξει κανείς δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Τώρα, αν δείτε τις, ε, τις εργα... τις μη εργάσιμες μέρες φτάνουμε σε 108. Και αυτό δεν είναι σωστό. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις ε, ελεύθερες ημέρες κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα έχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα δημόσια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν τροπολογίες που λέω σε αυτές τις ελεύθερες ημέρες να υπάρξει κάποια μετεκπαίδευση για να εξοικονομηθούν και οι δαπάνες και έχω καταθέσει και μια ε, συγκεκριμένη τροπολογία στο μέλλον προτείνω ε, business εισιτήρια θα πληρώνονται μόνο εάν ε, το ταξίδι ξεπερνάει τις 8 ώρες και ε, κατά τα άλλα οι διπλωμάτες να σας πω ότι δεν παίρνουν ποτέ ταξίδι εισιτήριο business. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καταθέσει τροπολογής για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων και revolving doors. Όμως κάτι θα κάνω και εκεί. Ε, έχω φτάσει σχεδόν στους ε, πληροφοριοδότες. Υπήρξε μία ακρόαση. Οι μένοι είπαν ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρη. Έχω, είμαι σε επαφή με τον διαμεσολαβητή και πρέπει να σου πω ότι είναι δύσκολο όμως να γίνει κάτι για αυτούς. Ε, αυτό που βρίσκω πολύ καλό στο σχέδιο της Κομισιόν είναι ότι στο μέλλον, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα υπάρχει ένα μητρό όπου θα αναφέρεται η εφαρμογή του καταστατικού στους διάφορους θεσμούς, δηλαδή όλες οι εφαρμοστικές πράξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να αποκτήσει κανείς μια γενική εικόνα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται το καταστατικό με τον ίδιο τρόπο παντού, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό äh, ευχαριστήσω την, εισηγήτρη. Ο κύριος Έρενχάουζερ ζητάει το λόγο και η κυρία Αγιάλα Σέντερ και μετά ο κύριος Μούλτερ, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νόμιζα ότι θα μιλάγε πρώτα ο κύριος Έρενχάουζερ. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πόσο, με πόση λεπτομέρεια δουλεύει η συγκήτρια. Και βέβαια και προσπαθεί να πετύχει και να πάει ακόμα πιο μακριά τους στόχου της έκθεσης αυτής. Η έκθεση αυτή όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια έκθεση πάρα πολύ λεπτή, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την βούλησή μας, Υπάρχει βούληση, αλλά υπάρχουν και δικαιώματα. Οι κοινωνικοί εταίροι και αυτοί έχουν κάτι να πούν. Δεν ε, πρόκειται για κάποιους οι οποίοι παίρνουν μόνο εντολές. Είναι ενεργά άτομα, οπότε φαντάζομαι ότι συζήτησε με τους κοινωνικούς εταίρους η συγκήτρια για όλα αυτά και ότι αντιλαμβάνεται πως υπάρχει ε, επιθυμία να προχωρήσουν αυτά. Τώρα, η σύγκριση που κάνει με Γερμανούς, για παράδειγμα, διπλωμάτες, δεν ξέρω αν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν είναι συγκρίσιμες ε, οι περιπτώσεις. Πάντως να υπενθυμίσω ότι το 2004 είχαμε μια τεράστια μεταρρύθμιση, ακόμα και πριν την ζητήσουμε εμείς όπως το είπε ίδια. Μεταρρύθμιση λοιπόν γενικού χαρακτήρα που έφτασε στη ρίζα της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης με μείωση 8 δις ευρώ μέχρι το 2020. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι τότε βρισκόμασταν σε μία περίοδο όπου προχωρούσαμε σε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 5.000 υπαλλήλους που είναι πολύ λιγότερο από ορισμένου δήμου στην Ευρώπη που γνωρίζουμε όλοι εδώ γιατί το έχουμε πει και ξαναπεί πολλές φορές. Ε, από εκεί λοιπόν αυξηθήκαμε και φτάσαμε πάνω από 500.000 ε, κάτι το οποίο το γνωρίζουν και όλοι μια που μπήκανε και άλλες χώρες και άλλοι πολίτες άλλων χωρών. Συνεπώς, εδώ, το θέμα δεν είναι να κόψουμε μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί. Το θέμα είναι να υπάρχει συνένεση με όλους εκείνους που από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο έκαναν την προσπάθεια αυτή το 2004 και έδειξαν αλληλεγγύη. Τώρα, πολύ συγκεκριμένα. Και εδώ νομίζω ότι η κυρία Ροντβέρνερ που ήταν αρχικά εισηγήτρια προσπαθεί να προχωρήσει σε μια νέα μεθοδολογία για υπολογισμό των συνταξιοδοτήσεων και προχωράει και σε ένα σύστημα αλληλεγγύης χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε εδώ. Μερικές τροπολογίες έτσι και αλλιώς απορρίφθηκαν ε, παλιότερα από την Επιτροπή μας και από ολόκληρο το Κοινοβούλιο όπως εκείνη η οποία λέει να μην προσλαμβάνουμε άτομα τα οποία έχουν απασχοληθεί στις μυστικές υπηρεσίες, δεν ξέρω εγώ ποιας χώρας. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια διάκριση και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να βάζουμε τέτοια ζητήματα εδώ. Έπειτα το θέμα των διακοπών ή το θέμα των ε, αδειών για επιμόρφωση, για ανάπαυση, το θέμα του να συγκρίνουμε τις διακοπές του ενός και του άλλου, ενώ όταν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό κάναμε τα τελευταία χρόνια και σε περίοδο κρίσης, έχουμε προβλήματα για να βρούμε και να προσλάβουμε καλούς υπαλλήλους για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Δίκηση. Συνεπώς, ένας υπάλληλος πρέπει να ε, προτιμήσει να έρθει εδώ από οπουδήποτε αλλού. Το θέμα του εκπατρισμού, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μας κάνουν να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία πραγματικά απαιτούνται ως περικοπές και όχι να κόβουμε μέρες ανάπαυσης ή να κόβουμε εισιτήρια για ταξίδια μπορεί να είναι 8 ώρες. Νομίζω ότι οι 8 ώρες που λέμε για να αυξηθεί το ωράριο εργασίας, ότι είναι υπερβολικό γιατί είναι πάρα πολύ. Ο καθένας μας κάνει μια ιδιαίτερη δουλειά εδώ. Οπότε μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα, 8 ώρου κάθε μέρα, Εμεί ήμασταν με υπαλλήλου στην Ικαράουα, στη Μαυριτανία, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλέ ώρε μερικέ φορέ, οι οποίοι βάζουν τον εαυτό του σε κίνδυνο βρισκόμενοι σε τέτοια μέρη. Προφανώ και απαιτούν κάποιε μέρε ανάπαυση ή να μπορούν να ταξιδεύουν κάτω από καλέ συνθήκε. Όλα αυτά ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να τα κόψουμε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να προσλαμβάνουμε του καλύτερου. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Άρα όπως συμβαίνει και με τη δημόσια δίκηση. Υπάρχουν κάποια προνόμια για τις διπλωματικές υπηρεσίες της χώρας μας και κάτι αντίστοιχο πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και εμείς για τους δικούς μας υπαλλήλου, να μπορούμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν. Για αλλιώ θα προσλαμβάνουμε τους χειρότερους και θα περιορίσουμε πάρα πολύ τη δράση μας και τις ικανότητές μας. Γι' αυτό πρέπει να περιορίσουμε τις ε, περικοπές στην αλληλεγγύη και στις συντάξεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και όχι να τη χειροτερέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γκρέσλερ, έχετε την ε, υποστήριξή μου για την ε, αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Υπάρχει μια τροπολογία που την έχετε ίσως διατυπώσει πιο με μεγαλύτερη οξύτητα από ότι εγώ. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει τώρα εμένα ιδιαίτερα είναι σημαντικό αν η Επιτροπή μας λαμβάνει υπόψη το θέμα της ε, αντιμετώπισης της διαφθοράς να λάβει υπόψη τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα για την προστασία των whistleblowers. Είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι το άρθρο 202α, 220β και γι' αυτό εμείς έχουμε μελετήσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και έχουμε διατυπώσει και τις συστάσεις αυτής της μελέτης σε τροπολογίες έχω μοιράσει αυτές τις, έχω διανύμει αυτές τις τροπολογίες, πρόκειται για 17 τροπολογίες. Δεν πρόκειται μονάχα για την προστασία των whistleblowers, πρόκειται για την προστασία των ε, ίδιων των θεσμικών οργάνων για να, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για να ε, κυλιδώσουν την αξιοπιστία των ηγετικών στελεχών σε σχέση λοιπόν με τη διαδικασία, σε σχέση με τι προθεσμίε, σε σχέση με τα δικαιώματα ακρόαση και όλα αυτά. Υπάρχουν πολλέ προτάσει που έχουμε καταθέσει για του whistleblowers, για αυτού οι οποίοι καταγγέλνουν κάτι. Και αν υπάρχουν και περαιτέρω προτάσει για βελτίωση, και αυτό πάντα μπορεί να ισχύει, θα είμαστε έτοιμοι να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα θα καταθέσουμε από τη δική μας πλευρά αυτές τις τροπολογίες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας και είμαστε απόλυτα στην διάθεση των πολιτικών ομάδων οι οποίες θέλουν και αυτές να παίξουν κάποιο ρόλο στη διατύπωση αυτών των προτάσεων. Ε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά την ε, διαφθορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την μοναδική μάλλον ευκαιρία σε αυτή τη δεκαετία για να ενσωματωθεί και αυτό το θέμα μέσα στο καταστατικό των υπαλλήλων και δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Κύριος Μούλτερ. Πολύ σύντομα, πρόεδρε. Εδώ πέρα πρέπει να δηλώσω ε, ενδιαφέρον ότι ήμουνα υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται να πάρω σύνταξη. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό προκαταλαμβάνει αυτά που θα πω. Έχω πάντως να κάνω δύο παρατηρήσεις προς την κυρία Δέσλερ. Πρώτα απ' όλα, το επίπεδο των ε, αμοιβών. Λόγος για τον οποίο ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, υπάρχει υψηλή αμοιβή είναι γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε υπαλλήλου γιατί έπρεπε να απομακρυνθούν από τις χώρες τους και το ίδιο ισχύει και για τις πρεσβείες, τις μόνιμες αντιπροσωπείες δηλαδή των χωρών μελών. Και εκεί πληρώνονται πιο υψηλή μισθή από ότι στους υπαλλήλου τους που βρίσκονται στις χώρες τους. Τώρα είναι δύσκολο να συγκρίνουμε ποιος είναι ο μέσος όρος μισθού ενός Γερμανού που δουλεύει σε μία μόνιμη αντιπροσωπεία. Πώς θα συγκρίνουμε αυτό με έναν υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να γνωρίζω ότι μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση Ξέρω μάλλον ότι μετά την τελευταία μεταρρύθμιση οι αμοιβέ δεν είναι τόσο ελκυστικέ. Και είναι αλήθεια. Θα έχουμε και την Κροατία τώρα. Ε, λοιπόν, σας προφορώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα διερμηνέα Κροάτη, γιατί οι αμοιβέ που τους δίνουμε είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με αυτά που μπορούν να κερδίσουν στις χώρες τους. Οπότε, τι είναι αυτά τα ποσά που συγκρίνουμε. Θα ήθελα να ξέρω, ώστε όταν κληθούμε να ψηφίσουμε, να γνωρίζουμε τι ακριβώς ψηφίζουμε. Όσον αφορά τις άδειε, τις αντιπροσωπείες κλπ. Και αυτό πρέπει να το συγκρίνουμε με τα κράτη-μέλη γιατί στις αντιπροσωπείες έχουμε και εθνικό προσωπικό, επιτόπου δηλαδή που το προσλαμβάνουμε, αλλά έχουμε και Ευρωπαίους ε, υπαλλήλους. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Εγώ δεν τις έχω δει ακόμα, εκτός αν μου έχουν ξεφύγει, αλλά θα ήθελα να τις έχω πριν ψηφίσω. Πρόεδρος, πέντε λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα θα έχουμε διερμηνία. Η κυρία Μακοβά έχει ζητήσει το λόγο και μετά νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε με την κυρία Κρέσλερ, τελευταία ομιλήτρια. Η κυρία Μακοβέ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο θέμα της δήλωσης συμφερόντων. Και ιδιαίτερα για την περίοδο του cooling off. Συμφωνώ ότι χρειάζεται υψηλή προστασία των whistleblowers, αυτών που αποκαλύπτουν δηλαδή πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πληροφορίες μέσα από τα θεσμικά όργανα γιατί ό,τι παρατυπίες γίνονται. Τώρα όσον αφορά τα ταξίδια σε business. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι πολύ κακό και αντιβαίνει σε κάθε είδου κοινή λογική να βλέπουμε σε περίοδο τέτοιας κρίσης ανθρώπους να ταξιδεύουν με business. Και βέβαια είμαστε και εμείς, αλλά τώρα μιλάμε για το προσωπικό. Συνεπώς στηρίζω απόλυτα τις διατάξεις αυτές που προτείνονται. Το ρώσο για τις ώρες εργασίας μάλλον ε, για το, τη θέση business στα ταξίδια να μην υπάρχει καθόλου. Τώρα ήμουνα στη Μολδαβία πριν από δύο μήνε και εγώ ταξίδεψα με οικόνομη, σε οικονομική θέση, γιατί έτσι θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω. Και το προσωπικό ταξίδευε σε business. Και μιλάμε για δύο πτήσει, έτσι. Ε, Βρυξέλλε βγαίνει και βγαίνει Κίσλοκ. Εμείς συζητούμε από τους συμπολίτες μας, στις χώρες μας, να δεχθούν μέτρα λιτότητας χαμηλότερους μισθούς, οι συντάξεις. Και γενικά του ζητάμε να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες ζωής. Και συγχρόνως δεν κάνουμε τίποτα για να μειώσουμε τις δικές μας τις δαπάνες. Πρέπει να μειώσουμε τις δικές μας τις δαπάνες. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο εξοικονομήστε, περιορίστε τις δαπάνες σας και εμείς να μην περιορίζουμε τίποτα. Για παράδειγμα τα ταξίδια αυτά που κάνουμε σε business και δεν αλλάζουμε τίποτα, ακόμα θέλουμε να αυξήσουμε και τον προπολογισμό, που αυτό βλέπω ότι γίνεται σε πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλε. Είπα ότι αυτό είναι ένα συγκινησιακό θέμα. Αλλά παρακαλώ να μην αναγνώρισετε σε αυτά που γράφω κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται. Δεν μίλησα για μισθού, μονάχα σε σχέση με το αν θα πρέπει να περιλαμβάνεται κάτι όταν και μήπως κάποιος ο οποίος έχει 10.000 ευρώ ήδη καθαρά, αν θα πρέπει να έχει επιπλέον και τόσο ελεύθερο χρόνο. Αυτό δεν είναι εύκολο να το αιτιολογήσουμε προς τον έξω κόσμο. Δεν έχω θίξει λοιπόν καθόλου το θέμα των αποδοχών των υπαλλήλων, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο εισόδου στο, σε επίπεδο μισθών, δηλαδή σε πάρα πολλά ε, επαγγέλματα. Και εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί σε επίπεδα πάνω από το βαθμό εισόδου, δηλαδή σε άντε 7 ή άντε 8. Επίσης έχουμε και την, ε, το επίδομα εκπατρισμού που είναι 16%. Δεν είναι η ίδια κατάσταση όπως την ε, διπλωματική αντιπροσωπεία των κρατών μελών που αλλάζουν τοποθέτηση τα, οι διπλωμάτες κάθε τρία χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί αυτή η αποζημίωση εκπατρισμού όταν έρχεται κανείς στις Βρυξέλλες και μένει για πολύ καιρό πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πάντα τους καλύτερους. Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτά που λέει ο κύριος Μούλτερ ότι έχουν ξεκινήσει Τώρα τα προγράμματα πούμε, για τους Κροάτες έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδεύσεις για τους ε, διερμηνείς από την Κροατία. Αλλά θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει η εκπαίδευση και να έχουμε αρκετούς διερμηνείς από, την, από τα κροατικά. Αυτό το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και με άλλες ε, γλώσσες, με τα σλοβάκικα και κτλ. Είναι πάντα ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε στους ε, ε, στις εντάξεις των χωρών αυτών και για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων και δεν συνδέεται με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Αν δεν κάνουμε τίποτα, τότε δίνουμε ένα θαυμάσιο πρόσχημα στους αντιευρωπαίους να μας επιτεθούν. Εγώ δεν έχω καμία ψευδέστηση για τα θέματα αυτά. Επομένως, οι προτάσεις αυτές εδώ πέρα που περιλαμβάνονται είναι ιδιαίτερα μετριοπαθείς. Ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι στην νομική επιτροπή δεν το βλέπουν με τέτοιο πνεύμα αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τα θέματα των ομάδων πιέσεως, των λόμπι. Παίρνουμε πάντα πάρα πολύ αρνητικά email, ξέρω πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, εγώ δεν το παίρνω πια προσεκτικά, προσωπικά συγγνώμη. Θέλω να έχουμε μια δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να λειτουργεί προ όφελο όλη τη Ευρώπη. Εγώ βλέποντα την διοίκηση των ευρωπαϊκών οργάνων όπω έχει σήμερα πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Θεωρώ ότι οι προτάσει μου είναι μετριοπαθεί και περιορισμένε. Πιστεύω ότι όλε αυτέ οι προτάσει θα πρέπει να συζητηθούν γιατί έχουν υπάρξει τεράστιες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών, όχι μονάχα λόγω της οικονομικής κρίσης. Αλλά και αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τους βουλευτές. Είναι καιρός να τα κάνουμε και για τους υπαλλήλους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έτσι έχει κλείσει και η συζήτηση για αυτό το σημαντικό σημείο. Κλείνω αυτό το σημείο και κλείνω επίσης και την συνεδρίαση αύριο στις 9 η ώρα και πάλι με την αυγούρα θα είμαστε εδώ.